Dear colleagues, I would like to suggest that we start the meeting uh, because we have a very long agenda today and I would like to start the meeting with the... Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συνεδρίαση με το 8 της ημερησίας διάταξης. Θα ήθελα εγκάρδια να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, τον κύριο Βαντεμπράντε, θα του δώσω αμέσως το λόγο γιατί ήρθε να να μας μεταφέρει τα αποτελέσματα μιας πολύ σημαντικής έρευνας την οποία έκανε σχετικά με το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής. Ο Λουκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητή Ντανούτα και αγαπητά μέλη της Επιτροπής. Ε, με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόσκλησή σας να σας παρουσιάσω ή να υπογραμμίσω αν θέλετε κάποια τμήματα της μελέτης της Επιτροπής των Περιφερειών ε, για την τοπική διακυβέρνηση. Η συνθήκη της Λισαβόνας τίθεται σε λειτουργία 8 χρόνια μετά από τις πρώτες θεσμικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό ε, γίγνεσθε σε επίπεδο θεσμικό. Υπάρχει αύξηση των αρμοδιοτήτων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι αρμοδιότητες οι οποίες θα βοηθήσουν την ε, μεγέθυνση της πολιτικής διάστασης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουμε σε μια πιο σταθερή πλέον θεσμική φάση και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε And our major role uh, now is to provide with the tools for implementing the treaty. We believe that the multilateral government Νομίζουμε ότι η πολύπλευρη αυτή, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι ένα πολύτιμο μέσο και σαν πολιτική όλοι αντιμετωπίζουμε ένα παράδοξο. Υπάρχουν πολλά παράδοξα βέβαια, αλλά αυτό το εντοπίζουμε κάπως πιο εύκολα. Όσο πιο ουσιαστική και σημαντική γίνεται η Ευρώπη στην καθημερινή ζωή των πολιτών της και σε επίπεδο νομοθετικό και σε επίπεδο επιρροής των στρατηγικών επιλογών, των εθνικών στρατηγικών επιλογών, τόσο περισσότερο περίπλοκη φαίνεται και απόμακρη από τις πραγματικές της ανάγκες. Η διακυβέρνηση είναι η λύση στην επιτυχή ευρωπαϊκή διαχείριση, αν θέλετε, της καθημερινότητας. Ιδιαίτερα λόγω ακριβώς της οικονομικής κρίσης, η ηγετική πολιτική τάξη, αν θέλετε, έχει προσπαθήσει να συγκεντρώσει στοιχεία για μια νέα συζήτηση. Αυτό φυσικά ισχύει και για τα μέλη, τα νέα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Περιφερειών. Όταν ξεκινήσαμε τη σύνταξη του εγγράφου μας τον προηγούμενο χρόνο, χτύπησε η κρίση και βιώσαμε τους τρεις πρώτους μήνες της οικονομικής κρίσης. Διαρωτήθημε λοιπόν για την ουσία αυτής της πρωτοβουλίας, τι νόημα θα είχε πλέον μετά από αυτές τις αλλαγές, και είδαμε ακριβώς ότι η παγκοσμιοποίηση εν πολλής αυξάνει το βάρος και τη σημασία του ρόλου της πολυεπίπεδης αυτής διακυβερνητικής δράσης. Οι οικονομικές ε, και χρηματοοικονομικές μάλλον και χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και σε επίπεδο τοπικό και περιφερειακό ε, μπορεί να γίνει στόχος, μπορούν να γίνουν στόχος ε, μέτρων και αποφάσεων και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο εθνικό. Έχει σημασία να κατανοήσει κανείς σε την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Η κάθετη διάσταση καλύπτει όλα τα επίπεδα της πολιτικής λήψης αποφάσεων από το σφαιρικό στο τοπικό και από το τοπικό στο σφαιρικό. Υπογραμμίζει την σταθερή σύνδεση ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική πολιτική και στην ενίσχυση, ανάγκη ενίσχυσης μάλλον της Ευρώπης και σύγκλησης. Όταν εφαρμόζει κανείς μία εκ των προτέρων συμπεφωνημένη στρατηγική, όπως ακριβώς τη στρατηγική για την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών κτλ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι και σε ιδιωτικό επίπεδο και σε δημόσιο επίπεδο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τις ευθύνε που έχει πλέον μια δημοκρατική κοινωνία. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση μπορεί να προσφέρει περισσότερα επίπεδα λειτουργικής συνεργασίας. Πρέπει να διευκρινίσω εδώ ότι δεν μιλάμε για μια νέα θυσμική συζήτηση, δεν μιλάμε για μια νέα δημιουργία οργάνων. Πάρα πολλοί έχουν υποφέρει στο παρελθόν από τέτοιου είδους συζητήσεις. Όπως είπα στην αρχή της ομιλίας μου, 8 χρόνια περιμέναμε να φτάσουμε στο σημείο το σημερινό και δεν θέλουμε να ξανανοίξουμε μια συζήτηση γύρω από τα θεσμικά, αλλά μια μορφή θεσμικής λειτουργικής συνεργασίας που θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τους στόχους μας, τους κοινούς στόχους. Αυτό θα διασφαλίσει μια νέα δυναμική στην ευρωπαϊκή πολιτική, μια ουσιαστική εταιρική σχέση ανάμεσα σε όλα τα επίπεδα, την λεγόμενη κάθετη επικουρικότητα, δηλαδή συμπεριλαμβάνοντας τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο οριζόντιας αλληλεγγύης και επικουρικότητας. Έχουμε λοιπόν εδώ μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση αλλά και μια ε, διακυβέρνηση με πολλούς πρωταγωνιστές και εμπλεκομένους. Αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, το θέμα είναι να δούμε ποιες είναι οι κοινέ αρμοδιότητες και όχι οι διαιρεμένες αρμοδιότητες. Η στόχοι η πολιτική της Ένωσης είναι κοινή πρέπει να ενισχύσουμε την κοινοτική δράση στους τομείς που βρίσκονται στην καρδιά θα έλεγα των ανησυχιών του Ευρωπαίου πολίτη. Οι συστάσεις της Λευκής Βίβλου υπογραμμίζουν τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οδηγηθεί σε μια πρακτική θα έλεγα δυνατότητα άσκηση της πολιτικής που να καλύπτει και τις τοπικές ανάγκες ακόμα και στα πλαίσια της εφαρμογής συνολικών κοινοτικών πολιτικών. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρυνθούμε και από το δικό σας επίπεδο στην, ε, ε, στην προσπάθειά μας αυτή. Εσείς ε, στα πλαίσια αυτά έχετε δημοσιεύσει ένα έγγραφο και ζητάτε από την Επιτροπή των Περιφερειών να συντονίσει τις προσπάθειές του καλύτερα και σε ποιοτικό και σε ποσοτικό επίπεδο. Και όπως είχαμε συμφωνήσει και με τον πρόεδρο Μπαρόσο, θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε συζητήσεις έτσι ώστε τους επόμενους μήνες ε, να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στην ε, μελλοντική ομάδα των επιτρόπων για τον τρόπο με τον οποίο καλύτερα θα γίνει σεβαστό και θα ακολουθηθεί το κείμενο το οποίο, βρίσκεται, το οποίο αντιπροσωπεύεται θα έλεγα από την ε, λευκή μας βίβλο. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης, η ενίσχυση της κοινοτικής διάστασης που είναι η καρδιά θα έλεγα της πολυεπίπεδης αυτής διακυβέρνησης. Απαιτείται λοιπόν ε, νομιμότητα σε επίπεδο λήψης αποφάσεων φυσικά αλλά και αποτελεσματικότητα πρακτική και μπορούμε να τα εγγυηθούμε αυτά εφόσον οι τοπικοί εταιροί, οι τοπικές αρχές είναι ουσιαστικοί πρωταγωνιστές και όχι τυπικοί συμμετέχοντες. Ακριβώς λοιπόν θα πρέπει να μπορούν να επηρεάζουν από κάτω προς τα πάνω η τοπική και περιφερειακή εταίροι τη λήψη αποφάσεων. Κάθε μεταρρύθμιση, μείζων μεταρρύθμιση ευρωπαϊκή θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα δράσης σε τοπικό επίπεδο, το οποίο θα περιλαμβάνει μια πολιτική δομή διευκόλυνσης της εφαρμογής και αξιολόγησης των εφαρμόσιμων πολιτικών. Αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και μια σωστή πολιτική ενημέρωσης. Συστήνουμε ολοκληρωμένες πολιτικές με σωστό συντονισμό ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και ουσιαστική εφαρμογή τομεακών πολιτικών έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνέργειες ανάμεσα στου εταίρους. Πίσω από κλειστέ πόρτες και σε διαδρόμους δεν είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών. Ζητάμε λοιπόν από κοντά εμπλοκή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαδικασία ε, λήψεως νομοθετικών αποφάσεων και στην αποκατάσταση των εσωτερικών ισορροπιών που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες αυτές. Υπογραμμίζουμε την σημασία που έχει η συστηματική χρήση των αναλύσεων περιφερειακών συνεπειών, των μεγαλύτερων μηχανισμών πολιτικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται και να εφαρμόζονται στο καταλληλότερο κάθε φορά επίπεδο υπό το φως των βασικών αρχών της επικορικότητας και της αναλογικότητας. Συστήνουμε παράλληλα καινοτόμες και καινοτόμες και συμμετοχικές πολιτικές διακυβέρνησης και πειραματισμούς σαν παράδειγμα ε, με τριμερείς συμβάσεις οι οποίες θα μπορέσουν να ενισχύσουν τις δυνατότητες περιφερειακής συνεργασίας από σύμβαση σε σύμβαση, από συμβόλαιο σε συμβόλαιο. Και θα συνεχίσω, λέει ο Βάντεν Μπράντε, στην Ολλανδική. Αγαπητοί φίλοι, Αγαπητοί Πρόεδρε, με τη θέση σε ισχύ λοιπόν της συνθήκης της Λισαβόνας θα πρέπει να αποφύγουμε να ξεκινήσει μια συζήτηση από την αρχή. Έχω την εντύπωση ότι η συζήτηση γύρω από τα θεσμικά προβλήματα θα πρέπει να γίνει πιο πρακτική σε επίπεδο διακυβέρνησης. Ο τρόπος με τον οποίο θα διακυβερνηθεί από εδώ και πέρα η Ευρώπη είναι το ζητούμενο. Η διαθεσμική συνεργασία είναι δεδομένη, η συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία λήψης απόφασης είναι μια ερώτηση η οποία κατά τη διάρκεια της επόμενης πενταετίας δεν θα πρέπει να αποφευθεί η συζήτησή της. Είναι καθοριστικές ερωτήσεις για την επιτυχία της κοινή στρατηγικής και την κοινή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Η νέα Επιτροπή έχει να αναλάβει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της ευθύνης και οι ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων στις αρχές του μηνός Ιανουαρίου θα είναι καθοριστική. Το θέμα βέβαια είναι να προσπαθήσουμε να δούμε σε ποιο σημείο θα φτάσουν οι νέες φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και γι' αυτό κυρία Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων εδώ ε, για την πρόσκλησή σας στις ακροάσεις αυτές και ε, σας συγχαίρω για την αντίληψη η οποία σας χαρακτηρίζει. Σχετικά λοιπόν με τη συμμετοχή μας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πρέπει να ενισχυθεί γιατί αυτό θα βοηθήσει την Ένωση να γίνει πιο αποτελεσματική. Οι συστάσεις της Επιτροπής Περιφερειών δεν έχει μόνο σαν στόχο την καλύτερη και αντιπροσωπευτικότερη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, αλλά έχει σαν στόχο την σαφή βελτίωση των εταίρων στα διάφορα επίπεδα των πολιτικών εταίρων, κάτι το οποίο θα προωθήσει και την κουλτούρα, αν θέλετε, της συνεργασίας. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής διαπιστώνοντας ότι ο Γέρζι Μπούζεκ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήρθε μας μίλησε και μας στήριξε στην τελευταία μας ολομέλεια τον προηγούμενο μήνα. Η συζήτηση γύρω από τα ευρωπαϊκά θέματα θα πρέπει να υπογραμμίζει κυρίως τα πολιτικά προβλήματα πλέον και όχι τα θεσμικά και συνταγματικά. Διαπιστώνουμε ένα παράδοξο. Οι θεσμοί ναι μεν αναζητούν και στοχεύουν την συνένεση, αλλά αυτή η συνένεση με τη σειρά της δεν έχει διευκολύνει όσο θα έπρεπε τουλάχιστον την πολιτικοποίηση με δημοκρατικό τρόπο της συζήτησης γύρω από τα ευρωπαϊκά θέματα. Αυτό ακριβώς εξηγεί τον λόγο για τον οποίο οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο που ζούμε σήμερα, έχει την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ζει και δεν τον ρόλο της ε, πλήρως. Το θέμα λοιπόν η συζήτηση είναι να γίνει πολιτική, γιατί τότε μόνο ο πολίτης θα κατανοήσει ότι τον ενδιαφέρει η συζήτηση αυτή γύρω από τα ευρωπαϊκά θέματα. Έχουμε εδώ να κάνουμε με μια αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει μια αδυναμία οι περιφερειακοί, τοπικοί εταίροι στα πλαίσια της εντολής τους θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους έτσι ώστε να προσπαθήσουν να συνεισφέρουν στην λύση των προβλημάτων που βιώνει ο Ευρωπαίος πολίτης. Η Λευκή Βίβλος είναι μια σαφής ελπίζω συμβολή της Επιτροπής των Περιφερειών στην κοινοτική ατζέντα σε εισαγωγικά. Πρόκειται για μια λευκή βίβλο η οποία δημοσιεύεται σε μια κομβική στιγμή της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους επόμενους μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να καταλήξει σε μια στρατηγική για την αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων όπως οι κλιματολογικές αλλαγές, η γύρανση του πληθυσμού του ευρωπαϊκού και οι συνέπειες που προκαλεί μια τέτοια, ένα τέτοιο φαινόμενο, και τα μέτρα τα οποία θα διασφαλίσουν μια συνέχεια και σταθερότητα ε, στην προσπάθεια ανάκαμψης οικονομικής που έχει ήδη ίσως ξεκινήσει. Όλα αυτά δείχνουν ότι θα πρέπει να επανέλθουμε και να προσαρμόσουμε τις μεθόδους διακυβέρνησης επί τη βάση των νέων μέσων που μας δίδει η Λισαβόνα. Η δυνατότητα πολιτικής πρωτοβουλίας πολιτών που δίδει η συνθήκη ξέρετε ότι ε, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποβεί Υπάρχει ε, μια μεγάλη ομάδα δημάρχων και ε, γενικά ερετών αντιπροσώπων από τις διάφορες χώρες της Ευρώπης που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το μέσο αυτό. Άλλο παράδειγμα, την επόμενη εβδομάδα στην Κοπενχάγη θα υπάρξει μια παγκόσμια διάσκεψη η οποία θα φέρει σε επαφή χιλιάδες δημάρχους και τοπικούς άρχοντες από όλες τις χώρες του κόσμου και φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για επίπεδα δηλαδή συνεργασίας τα οποία είναι αποσυγκεντρωτικού τύπου, είναι επίπεδα συνεργασίας σε εντελώς περιφερειακό επίπεδο και θα συνεισφέρουν αυτά τα επίπεδα συνεργασίας στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως οι κλιματολογικές αλλαγές και οι συνέπειές τους. Υπάρχουν και άλλα φόρα τα οποία θα είναι χρήσιμα όπως η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη. Αυτές τις μέρες προετοιμάζουμε την συνάντηση των τοπικών και περιφερειακών αρχών των μεσογειακών περιοχών και υπάρχουν γενικότερα πολλά παραδείγματα και πολλά επίπεδα δράσης κοινής. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι και η Περιφερειακή Επιτροπή θα παίξει το ρόλο της, να δούμε ακριβώς τι θα γίνει και με τις λεγόμενες μακροπεριφέρειες και τη στρατηγική μας ε, την μακροπεριφερειακή, για παράδειγμα στις παραδουνάβιες περιοχές ή και στην Βαλτική. Και φυσικά εδώ δεν θα πρέπει να αγνοούμε και κάποιες ολοκληρωμένες πολιτικές όπως η πολιτική για τις θαλάσσιες μεταφορές ε, που επηρεάζει πάρα πολλές χώρες. Υπάρχουν ε, λοιπόν δυνατότητες και επίπεδα συνεργασίας. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το χρόνο έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει τον ρόλο τον οποίο μπορεί να παίξει και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να μεταφερθεί με σωστό τρόπο και προσαρμοσμένη στις τοπικές ανάγκες σε κάθε χώρα. Έχουμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον οποίον στόχος είναι να λάβουμε υπόψη μας μια δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης που θα συμπέσει και με τη δημοσίευση του νέου προγράμματος δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις αρχές του 2010. Θέλουμε να βοηθήσουμε επίσης τις εργασίες και της ομάδας, της λεγόμενης ομάδα των σοφών ή ομάδα των επαϊόντων, ε, ο πρόεδρος της ομάδας αυτής είναι ο Φελίπε Γκονσάλες και στόχος τους είναι να δουν πόσο οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Γίγνεσθε μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας οι οποίες τους παρέχονται σήμερα. Πρόκειται για κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει νέου τύπου θεσμικά επίπεδα λήψης απόφασης, αλλά πρόκειται για κάποιες νέες μορφές, άτυπης μερικές φορές, αλλά χρήσιμης πολύ συνεργασίας. Η ιδέα αυτή ελπίζουμε να γίνει δεκτή και από την πιο συγκεκριμένα από την ομάδα αυτή των επαϊόντων. Λοιπόν, ε, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά είναι τα κάποια πρώτα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν, αν θέλετε, την ουσία σε αδρές γραμμές βέβαια της Λευκής Βίβλου την οποία έχουμε συντάξει πρόσφατα. Έχω την εντύπωση ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου πως ε, και εσείς θα μπορέσετε να συνεισφέρετε και με κριτικό βλέμμα ή και να προτείνετε επίσης και διαφορετικές πορείες δράσης. Συνεχίζει στα γαλλικά ο Βάντεν Μπράντε. Αυτές οι πρωτοβουλίες, ε, οι δυνατότητες λαϊκής πρωτοβουλίας που δίνει η συνθήκη ελπίζω να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης και ελπίζω να χρησιμοποιηθούν. Είναι νέες προοπτικές, προοπτικές οι οποίες ανοίγουν μια νέα περίοδο θα έλεγα συνεργασίας και διαβούλευσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι εισερχόμαστε τώρα στη νέα φάση, στο νέο στάδιο της ε, συζήτησης ε, του πολιτικού θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτό το έγγραφο 2020 για το 2020 υπάρχουν σαφείς στόχοι αυτού του πολιτικού θεματολογίου τους οποίους συμμεριζόμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο της όλης συζήτησης και κέριο θέμα είναι το θέμα της διακυβέρνησης. Η συνεισφορά που ακούσαμε μόλις από την Επιτροπή Περιφερειών θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη για μας στην προσπάθεια περισυλλογής που θα κληθούμε να κάνουμε για το πώς θα επιτύχουμε τους στόχους του θεματολογίου αυτού. που είναι στόχοι και της περιφερειακής πολιτικής ευρύτερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ κύριε Πρόεδρε των, της Επιτροπής των Περιφερειών. Υπάρχει δυστυχώς ε, πίεση χρόνου. Στις 10 ακριβώς θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι της ε, συνεδριασής μας. Οπότε αν θέλετε να μιλήσετε θα πρέπει να το αποφασίσετε τώρα για να εγγραφείτε στον κατάλογο. Ο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε για την ε, ενημέρωση τον κύριο Μπράντε. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Φαίνεται πως από έρευνα του Ευρωβαρόμετρου φετινή το 50% των Ευρωπαίων πολιτών εμπιστεύονται περισσότερο τους περιφερειακούς και τοπικούς εκπροσώπους σε σχέση με την κυβέρνηση της χώρας τους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα στην ίδια έρευνα ε, βλέπω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες εκτιμούν ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές το 59% των ε, Ευρωπαίων πολιτών εκτιμά ότι δεν παίρνονται υπόψη στην ευρωπαϊκή διαδικασία. Ήδη βλέπουμε ότι αναβαθμίζεται ε, σε σχέση με το παρελθόν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που θα δώσουν την απάντηση σε αυτούς τους Ευρωπαίους πολίτες ότι οι προσδοκίες τους μπορούν να επιβεβαιωθούν. Δηλαδή, στην πράξη και πέρα από τις καλές προθέσεις ή τα καλά, τα ωραία λόγια, πώς μπορεί να αναβαθμιστεί ο λόγος και η άποψη των ε, περιφερειακών και τοπικών αρχών. much. Λαμπέρ uh, Ευχαριστώ. Λαμπέρ Βανίστελ Ροϊ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είμαστε ευτυχείς που υποδεχόμαστε τον κύριο Βάντερ Μπραντ, πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών. Θεωρούμε ότι η ομιλία του ήταν πολύ σημαντική. Εντάσσεται σε μια συζήτηση που εμείς εδώ έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό και νομίζω ότι είναι ασφαλές να πει κανείς ότι στην πράξη όλα αυτά μπορούν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμα. Είναι δε αντικείμενο συζήτησης και σε επίπεδο κρατών μελών, συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και Ένωσης, περιφερειακών ε, οντοτήτων και Ένωσης και με τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, η κατάσταση δεν έχει ουσιαστικά αλλάξει. Η θέση των κρατών μελών δεν έχει αλλάξει. Το 70% των πρωτοβουλειών ε, λαμβάνεται ως απόφαση σε επίπεδο περιφερειών. Για την κλιματική μεταβολή είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα αμφισβητήσει κανείς ε, την στοχοθέτηση που προδιαγράφεται. Οπότε νομίζω ότι το θέμα είναι συνενετικό, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε, τι θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να κάνουμε αν τελικά δεν κινηθούν τα πράγματα με την ταχύτητα που προβλέπετε. Μιλάμε για την περιφερειακή συνοχή, είναι ένας νέος στόχος το έχετε σκεφτεί αυτό, σας έχει απασχολήσει ως Επιτροπή των Περιφερειών. Θεωρείτε ότι τώρα έχετε τη δυνατότητα να διαδραματίσετε ένα πολύ πιο ενεργό ρόλο. Θέλετε να διαδραματίσετε έναν πιο ενεργό ρόλο. Ούτως ώστε οι πολίτες να έχουν πραγματική δυνατότητα παρέμβασης στα διάφορα επίπεδα. Αυτή την συμμετοχική διαδικασία που αναφέρατε. Σας άκουσα κάπως ε, διστακτικό, μετριοπαθή. Θεωρείτε ότι αυτά που μας είπατε επαρκούν ή θα πρέπει να αυξήσουμε ενδεχομένως το επίπεδο φιλοδοξιών μας. Ευχαριστώ. Γιάννη Ολμπριχτ. Ε, Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca, chciałbym e, zwrócić uwagę na pewien element. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω ένα στοιχείο το οποίο είναι σχετικά επικίνδυνο. Οι συνθήκες όπως προκύπτουν μετά από την κρίση πάντα ευνοούν την εξαγγελία μέτρων υπέρ της αποτελεσματικότητος, της ανάκαμψης, της βελτίωσης των πραγμάτων. Ο κίνδυνος για τον οποίο νομιλούσα είναι να δημιουργηθεί μια ακόμα πιο κεντρική δομή και διαδικασία διαχείρισης για λόγους απλούστευσης και για λόγους ε, χρόνου, ότι οι αποφάσεις σε καιρό κρίσης πρέπει να λαμβάνονται επιγόντως, ταχαίως. Μήπως όμως πρόκειται για υπεραπλούστευση αυτοί που δρούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν περισσότερο, διότι είναι αποτελεσματικότερη η συνεισφορά τους στην επίλυση της κρίσεως. Τα πρόσφατα έγγραφα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν το διορισμό, πριν να αναλάβει ε, το νέο συλλογικό σώμα, αντανακλούν σαφώς, πιστεύω, την άποψη υπέρ της εξειδίκευσης και όχι του οριζόντιου χαρακτήρα. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός, μια τομεακή αν θέλετε προσέγγιση, η οποία μοιραία οδηγεί σε κεντρικής φύσεως δομή διαχείρισης. Τώρα κάτι άλλο η πολυτομεακή, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση θεωρείται από ορισμένους ως αναγκαιότητα για την διαχείριση και την επίτευξη των στόχων μας. Ο καθής να πράττει αυτό που του αναλογεί χωρίς να εμποδίζει το έργο του άλλου. Η Επιτροπή των Περιφερειών, και συγγνώμη που το λέω έτσι, μπορεί να θέλει να υιοθετήσει μια τέτοιου είδους προσέγγιση. Όμως η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση πιστεύω ότι δεν σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι ο καθένας στη γωνιά του κάνει κάτι χωρίς να επικοινωνεί με τον άλλον. Όχι. Αρμονική, αγαστή συνεργασία είναι αυτό που χρειάζεται. Συνεργασία και επικοινωνία και όχι στεγανοποίηση και κατακαιρματισμός των στόχων. Ευχαριστώ. Λουκ, μπορείς να σχολιάσεις. Ε, ε, ε. Κύριε Τρεμόπουλε, ορθά αναφερθήκατε στο Ευρωβαρόμετρο. Η Ρίστο Εμπαρόδο είναι η πρώτη φορά κατόπιν από έτοιμά μας που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενσωμάτωσε στο Ευρωβαρόμετρο πέντε ερωτήματα που αφορούν το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 50 χρόνια μας πήρε να συνειδητοποιήσουμε ως Ένωση την ανάγκη ότι που ε, να μεταφράσουμε με όρους ευρωβαρομέτρου τις ε, και ανησυχίες του πληθυσμού που ζει σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ή που διαχειρίζεται τα πράγματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Από την άλλη, λέτε ότι υπάρχει ένα 60% της κοινή γνώμης που αναφέρει ότι οι εκπρόσωποι του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου δεν κάνουν ό,τι θα μπορούσαν να κάνουν. Ε, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, διότι δεν έχουν πολλές φορές τη δυνατότητα να το κάνουν. Δεν έχουν τις αρμοδιότητες, την εξουσία να το κάνουν. Πάντως ουσιαστικά έχετε δίκιο. Ουσιαστικά έχετε δίκιο. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι πώς θα επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν λέγω ότι η προσέγγιση αυτή του, η πολυεπίπεδη θα αποτελέσει πανάκια, μαγικό ραβδί επίλυσης όλων των προβλημάτων. Όχι. Αλλά η μετανάστευση η αγορά απασχόλησης, το περιβάλλον, και θα επανέλθω από αυτό, πρέπει να περάσουν στη σφαίρα αρμοδιότητος του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου. Ο τοπικός όμως και περιφερειακός άρχον θα πρέπει να είναι και Ευρωπαίος άρχον. Και επ' αυτού πολλά ακόμα δεν έχουν γίνει. Είναι σημαντικό νομίζω να αναφέρουμε ότι πήραμε την πρωτοβουλία να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Όχι μόνο για να γνωρίσουμε σε, περισσότερο, σε μεγαλύτερο βάθος ε, τι συμβαίνει στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και για να οθήσουμε τους τοπικούς και περιφερειακούς άρχοντες να κινητοποιηθούν, να τους ε, διαφωτίσουμε για το τι πρέπει να γίνει ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε ούτως υπήν υπεργολάβοι κάποιων αποφάσεων που λαμβάνονται σε πιο κεντρικό επίπεδο. Οπότε υπάρχει προσδοκία. από τους πολίτες. Να δοθούν δυνατότητες και αρμοδιότητες στους άρχοντες του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου, αλλά συγχρόνως αυτοί να εμπλακούν περισσότερο στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Ένα παράδειγμα, όταν μιλούσα για επικοινωνία, ανέφερα την λευκή βίβλο όχι μόνο για τα σύμφωνα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά για μια απόφαση που θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα τοπικό ή περιφερειακό ε, προγραμματισμό και σχεδιασμό. Πάντα με εκπλήσει το γεγονός ότι πριν από δεκαετίες, όταν ταξιδεύαμε στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους, βλέπαμε ευχαριστούμε Ευρωπαϊκή Ένωση, ευχαριστούμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτός ο αυτοκινητόδρομος ε, θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά εξαφανίστηκαν, δεν υπάρχουν πια. Αποτελούν μια αναγνώριση των επιτυχιών μας. Κύριε Βανίστελ Σημειώνω την ε, παρατήρησή σας. Είναι κέρια, όντως. Εξάλλου η Επιτροπή Περιφερειών είναι ακόμα νέα. Πριν από 15 χρόνια συστάθηκε ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εόρτασε τα 50 χρόνια της γέννησής του. Βέβαια, στην αρχή ήταν εμβριακή η κατάσταση του με έξι κράτη-μέλη, τους λεγόμενους πατέρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ, μάθαμε πολλά, κατανομήσαμε ότι η Ευρώπη δεν οικοδομείται μόνο σε κεντρικό επίπεδο. Έχουμε προοδεύσει λοιπόν πολύ, αλλά πολλά ακόμα υπολείπονται. Και είναι μια καθημερινή μάχη αυτή που θα πρέπει να δώσουμε. Καθημερινή μάχη. Σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα μέτωπα. Και εγώ θα ήθελα να επανέλθω, μάλλον θα ήθελα να επανέλθω ε, εκ νέου ε, στο ερώτημα του κυρίου Τρεμόπουλου. Δώσαμε μάχη για να συνεργαστούμε με τα τοπικά, μάλλον με τα εθνικά ε, κοινοβούλια και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά αποτελούν πρόοδο και είναι απαραίτητα σήμερα. Κύριε Βανίστελ Ροϊ, Αναφέρατε το παράδειγμα της διάσκεψης για την κλιματική μεταβολή. Είχαμε τη δυνατότητα να, αναφέρουμε την άποψή μας στον κύριο Παρόζο, στον κύριο Πίμπαλξ, τον Επίτροπο για την ε, Ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικά για μας, διότι τα προβλήματα που αφορούν την κλιματική ε, μεταβολή κατά κύριο λόγο αφορούν όχι την Ήπεθρο, αλλά τα αστικά κέντρα. Η πυκνότητα του πληθυσμού, το κυκλοφοριακό, η ρήπανση, η πολεοδομία, οι εκπομπές ε, αερίων που συνεισφέρουν, τέλος πάντων συμβάλλουν στην δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς ε, είμαστε άμυροι ευθυνών ή ότι δεν θα πρέπει να ε, ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό και στο δικό μας επίπεδο. Η πρόκληση πάντως που θα χρηστεί να αντιμετωπίσουμε και αποτελεσματικά είναι να μην θέσουμε σε νέα βάση ή να μην θέσουμε εκ νέου το θεσμικό θέμα. Είχε ακουστεί ως και η ιδέα μιας ευρωπαϊκής γερουσίας ε, για την εκπροσώπηση σε περιφερειακό και ε, τοπικό επίπεδο. Εμείς δεν είμαστε υπέρ αυτής της λύσεως. Ξέρω ότι ορισμένοι ε, στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, το αντιμετωπίζουν ως ένα ευκταίο ενδεχόμενο. Πάντως ε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να θέσουμε σε νέα βάση το θεσμικό ζήτημα να μας απασχολήσει, να το σκεφτούμε, αλλά στα πλαίσια των υφισταμένων θεσμικών ε, κανόνων και αρμοδιοτήτων, των μεν και των δε. Είμαστε 27 σήμερα και δεν μπορούμε να περιπλέξουμε θεσμικά τα πράγματα. Η ανάλυση αντικτύπου. Η μελέτη αντικτύπου είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο. Να λάβουμε υπόψη μας δηλαδή, αλλά και να συγκεράσουμε συγχρόνως τις διαφορετικές απόψεις με στόχο την επίτευξη των κοινών στόχων. Εμείς ε, γύρω από αυτόν τον άξονα περισυλλογής έχουμε εργαστεί τους τελευταίους έξι μήνες. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι το οποίο βεβαίως είναι ε, κάτι που θα πρέπει να τονίσω. Τώρα, Αναφέρθηκε σε αρχικότερο στάδιο μια σειρά προσανατολισμών και θεωρήσαμε σε αυτό το στάδιο ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εμπειρία των ε, εκπροσώπων των ε, τοπικών και περιφερειακών αρχών. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας η Επιτροπή των Περιφερειών έχει σήμερα επίσημη δυνατότητα, αρμοδιότητα δηλαδή, να υποβάλει ε, συγκεκριμένες ε, προτάσεις, εκκλήσεις, συστάσεις και ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε αυτή τη νέα μας θεσμική θέση. Ας μην αυταπατώμεθα βεβαίως από την άλλη. Θα πρέπει ας πούμε να αναγνωρίσουμε ότι ο, κανείς δεν μπορεί να επηρεάσει ή να αλλάξει τον κόσμο μόνος του. Χρειάζεται συνεργασία. Συνεργασία στο εσωτερικό το δικό μας, στην Επιτροπή Περιφερειών, συνεργασία της Επιτροπής των Περιφερειών με τα λοιπά θεσμικά όργανα και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το πρωτόκολλο επικουρικότητος της ε, συνθήκης αναφέρει πολλά χρήσιμα στοιχεία για την συνεργασία αυτή. Στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αξιοποιήσουμε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η επικοινωνία με την Επιτροπή σας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα είναι εξαιρετικά σημαντική. Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συντάξουμε πιο πρακτικά έγγραφα τα οποία θα επηρεάσουν τα πράγματα. Δεν θα πρέπει δηλαδή να μπαίνουν, ε, να θάβονται ε, σε ένα σιρτάρι, όπως δυστυχώς συχνά γινόταν μέχρι τώρα. Και ελπίζω έτσι, στόχοθετημένα και συγκεκριμένα, να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Βεβαίως, υπάρχουν κίνδυνοι. Διότι οι προκλήσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές. Και αν δεν λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις με την, στον κατάλληλο χρονισμό, τα πράγματα θα επιδεινωθούν. χρόνος όμως είναι και μια ευκαιρία η κρίση. Εγώ ποτέ δεν μίλησα για μια εναλλακτική Ευρώπη, για δύο Ευρώπες αν θέλετε, για μια Ευρώπη των πόλεων και μια Ευρώπη των περιφερειών. Όχι, θα ήταν παράλογο αυτό. Η βάση της διακυβέρνησης είναι η ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων, των διαφοροποιήσεων των ε, διαφόρων επιπέδων και η κάλυψή τους στο σωστό επίπεδο με τα σωστά μέτρα. Υπάρχει η Επιτροπή Στόιμπερ που έχει ενσκύψει από αυτών των θεμάτων και που έχει συντάξει διάφορα έγγραφα, ας πούμε, για το στόχο της ε, μείωσης κατά 25% του διοικητικού άχθους. αν καταφέρουμε να μειώσουμε ε, το διοικητικό άκθος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί όμως να αποδειχθεί ότι αυξάνεται αυτό, το διοικητικό άκθος δηλαδή, σε εθνικό επίπεδο. Απευθύναμε επιστολή στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, περιφερειακή πολιτική και του επισημάναμε ότι αυτή η λογική στα άκρα της αντιβαίνει της όλης αρχής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, συνοχής και σταδιακής οικοδόμησης. μου είπε ο πρόεδρος ότι μιλάτε επί τη βάση ενός εγγράφου που δεν υπάρχει. Και εγώ του είπα, ναι, αυτό είναι το non-paper ένα έγγραφο που δεν υπάρχει. Και ως ε, Επιτροπή των ε, Περιφερειών, όντως θεσμικά μπορούμε να τοποθετηθούμε μόνο όταν υπάρχει μια ε, συγκεκριμένη πρόταση αλλά μπορούμε να πυροδοτήσουμε και τον ε, μηχανισμό της έγκαιρης προειδοποίησης. Διότι αν κινηθούμε προς μία τομεακή κατακαιρματισμένη πολιτική θα θέσουμε σε κίνδυνο, θα θέσουμε σε αμφισβήτηση τον ίδιο το στόχο της συνοχής και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στη Θουριγγία που είχα πάει πρόσφατα είδα μια έκθεση για τα πλεονεκτήματα της ε, πολιτικής συνοχής και ήταν ε, ε, σαφές το μήνυμα που ήθελε να περάσει η έκθεση, ότι υπέρ αυτού είμαστε. Συμμερίζομαι την άποψή σας, είναι και θέμα αξιοπιστίας. Αλλά δεν είναι δυνατόν να υιοθετήσουμε πολιτικές απομόνωσης πολιτικές άκρος τομιακές που θα μας απομονώσουν, που θα μας διχάσουν. Ο στόχος είναι γενικός, είναι οριζόντιος. και θα πρέπει να σκεφτούμε αυτή την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, αλλά εγώ θα μιλούσα πιο πολύ για διακυβέρνηση που περνάει από πολλούς φορείς. Και αυτά είναι σημαντικά να τα ξεκαθαρίσουμε τώρα, για να μην προκύψουν παρανοήσεις στο μέλλον. Είναι θέμα των πολιτικών που θα πρέπει να εφαρμόσουμε με τρόπο που να μας δώσει τη δυνατότητα να αποφύγουμε τον κεντρικό, το συγκεντρωτικό δηλαδή χαρακτήρα διακυβέρνησης. Και για να το επιτύχουμε αυτό χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων, μεταξύ των διαφόρων αρμοδίων στα διάφορα επίπεδα. Ναι. Ε, εδώ χρειάζεται μια υποστήριξη γιατί δεν, είναι, δεν πρόκειται εδώ για έναν αυτοσκοπό. Έχει υπάρξει ένα κενό στη συνθήκη του Μάστριχ το οποίο έπρεπε να πληρωθεί και πραγματικά αυτό είναι τεράστια σημασία για σας πως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε πλέον πολύ σημαντικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον προϋπολογισμό αλλά και άλλους τομείς. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας στηρίξετε επίσης. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε αυταπάτες βεβαίως όσον αφορά τον εχθρό μας, αν μου επιτρέπετε να το διατυπώσω έτσι. Από διοργανική άποψη, ωστόσο, έχουμε, είμαστε, συνεργαζόμαστε. Και μία πτυχή των διευρυμένων αρμοδιοτήτων που έχετε τώρα βάσει τις συνθήκες της Λισαβόνος και την οποία θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε από κοινού, ούτως ώστε να ασκήσουμε μια καλή πολιτική. Δύο ερωτήσεις. Ε, ο κύριος Μπλάσακ. Ναι, ε, σε σχέση με, τις, ε, με την χθεσινή ομιλία της, του Σώματος Συνέλευσης των Περιφερειών, αναφέρθηκε ο κ. Βάντερ Μπράντε στην παρουσίαση της Λευκής Βίβουλου ότι η βασική αρχή της σωστής διακυβέρνησης είναι πάντοτε η εταιρική σχέση και η συνεργασία. Η έρευνα δείχνει ότι η τοπική και περιφερειακή πολιτική έχουν τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πολιτών. Αλλά υπάρχουν άλλες έρευνες που δείχνουν ότι οι αντιπρόσωποι αυτοί, οι πολιτικοί αυτοί έχουν συχνά χαμηλό επίπεδο γνώσης όσον αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της και το τι μπορούν να κάνουν για τις ε, περιφέρειες και τις δημοτικές αρχές. Γι' αυτό θα ήθελα να υποστηρίξω την ιδέα ενός είδους εράσμους για τους ερετούς αντιπροσώπους, ιδέα την οποία παρουσίασε ο Ζαν Μαρί Πούπε στο προηγούμενο κοινοβούλιο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω το πώς θα υποστηρίζατε ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα και πώς θα εννοούσατε την εφαρμογή του στο εγγύς μέλλον. Ε, στο Κοινοβούλιο γίνεται η συζήτηση εν σχέση με, τις, ε, με το έργο της Επιτροπής των Περιφερειών και υπάρχουν διάφορες φωνές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι η Επιτροπή των Περιφερειών μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν διαφορετικό ρόλο. Και θα ήθελα να σας πω το εξή. Η δική μου βασική επιτροπή είναι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, όχι αυτή η αγορά. Και σε αυτή την, αγορά, ε, σε αυτή την ε, επιτροπή, συγγνώμη, ε, βάλαμε ε, στο τραπέζι τη συζήτηση για την καθυστέρηση των πληρωμών. Αυτή η οδηγία μεταχειρίζεται ε, διαφορετικά τους ιδιώτες από το δημόσιο. για ένα νοσοκομείο δηλαδή όταν υπάρχουν καθυστερήσεις θα πρέπει να πληρωθούν από την πρώτη μέρα επιτόκια. Κάτι το οποίο δεν ισχύει για τους ιδιώτες. Ε, δεν ξέρω γιατί ε, δεν γίνονται αντίστοιχα πράγματα στο τοπικό επίπεδο. Βλέπουμε πάντοτε η έρευνα επιπτώσεων στην Επιτροπή και αυτή τη φορά υπήρξε μια έρευνα επιπτώσεων όσον αφορά τον έλεγχο της επικουρικότητας. Και γιατί δεν διενεργείται πραγματικά ένα σωστό έλεγχο στο έγγραφό σας μιλάτε για τη δικτύωση μέσω του ίντερνετ. Αυτή θα ήταν μια δυνατότητα η Επιτροπή των Περιφερειών να βελτιώσει τη δικτύωση μέσω του ίντερνετ σε τοπικό επίπεδο. Γιατί το ερώτημα του τι μπορούμε να κάνουμε μετά τη Λισαβόνα, πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε περισσότερο την τοπική και περιφερειακή διάσταση, στην ερώτηση αυτή δεν έδωσε κανείς μέχρι τώρα μία απάντηση ο κύριος Κάντεκ και στη συνέχεια ο κύριος ε, Λάσακ. Θα κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Κάντεκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Απλώς θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για να σας υπενθυμίσω ότι αντιμετωπίζει κανείς έναν ε, περιφερικό οργανισμό διαφορετικά ανάλογα με τη χώρα και είναι οι χώρες αυτές ε, που αποφασίζουν για το επίπεδο κεντρικής οργάνωσης ή όχι. Υπάρχουν χώρες που είναι πιο, έχουν πιο κεντρική οργάνωση. Ε, η Γαλλία, για παράδειγμα, στη Γερμανία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν υπάρχει το ίδιο επίπεδο όσον αφορά τις αρμοδιότητες και δεν υπάρχει και η ίδια γεωγραφική οργάνωση. Λοιπόν, μπορούμε Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το στοιχείο της ποικιλία όσον αφορά την περιφερειακή οργάνωση. Και έστω και ε, και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε μια εναρμόνιση των περιφερειών στις διάφορες χώρες, παρόλο που αυτό μου φαίνεται πολύ δύσκολο, όπως είπα. Από την άλλη, νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε να μην ε, αντιταχθούμε σε αυτό το οποίο μας ενώνει, δηλαδή μια Ευρώπη των εθνών και μια να εντάξουμε μια Ευρώπη των εθνών σε μια Ευρώπη των περιφερειών. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό να μην το κάνουμε. Αλλά δεν θα πρέπει βεβαίω να παραβλέπουμε το ενδιαφέρον των περιφερειών και τη αποκέντρωση που επιτρέπει μια καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών ταμείων. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εδώ. Είμαστε η Ευρώπη των 27 εθνών και όχι των 27 περιφερειών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο. Καταρχήν θα ήθελα να συγχωρώ την Επιτροπή των Περιφερειών για τη σημασία αυτής της λευκής ε, βίβλου για τη διακυβέρνηση πολλαπλών επιπέδων. Και θα ήθελα να φερθώ στην συγκεκριμένη στρατηγική της Λισαβόνος. Ε, ε, ε, φαντάζομαι ότι έχει υλοποιηθεί το σχέδιο μεταρρύθμισης ε, έτσι όπως ε, βάσει των προτάσεων παρουσίασαν όλες οι χώρες. Η Κομισιόν θα καταρτήσει μια έκθεση για το Ερεινό Συμβούλιο. Θα ήθελα να σας πω πώς τοποθετήσετε έναντι τη στρατηγικής της Λισαβόνας και έναντι μιας νέας στρατηγικής. Ε, ποιες είναι οι βελτιώσεις που προπτήθησε να κάνετε από την άποψη της Επιτροπής των Περιφερειών. Ε, θα είμαι σύντομος. Κύριε Φλάσεκ, μια σωστή διακυβέρνηση, η χρηστή διακυβέρνηση βασίζεται σε εταιρικέ ε, σχέσεις και οι εταιρικέ σχέσεις σχετίζονται με τη σωστή διακυβέρνηση. Από το 2001 έχουμε τη Λευκή Βίβλο και τίθε το ζήτημα τη σωστή διακυβέρνηση και στην Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά υπάρχει, έχει ξεχαστεί λίγο η πρόταση της Επιτροπής της εποχής εκκίνησης. Θα πρέπει να της δώσουμε τώρα νέα ζωή. Βεβαίως είμαι υπέρ της πρότασης ενός εράσμους σε τοπικό επίπεδο, την ιδέα που παρουσίασε ο κ. Μποπή. Μπορώ να πω όταν, ότι όταν εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνετε τα κονδύλια για να γίνει κάτι τέτοιο, εγώ θα είμαι ο πρώτος εταίρος που θα συνεργαστεί μαζί σα. Δεν θέλω να σας ρίξω το παλάκι αλλά νομίζω ότι πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική ιδέα. Και σε μια δημοσίευση που αναφέρεται στη διακυβέρνηση πολλαπλών επιπέδων, τη Λευκή Βιβλία κλπ. Αναφέρουμε ρητά αυτή την ιδέα. Είναι κάτι που το εξετάζουμε τόσο ή Κυρία Ρούλε, ε, είναι προφανές ότι η ερώτηση αφορά να έχουμε μια πιο σωστή διακυβέρνηση, όχι μια περισσότερη διάσπαση. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε, προσπαθούμε να συστήσουμε το λεγόμενο δίκτυο επικουρικότητες και πάρα πολλές περιφέρειες συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο ανταλλάσσοντας όχι μόνο απόψεις αλλά και ε, παρουσιάζοντας κάποιες ιδέες ε, για νέες πολιτικές στις χώρες μέλη, κάτι το οποίο αναφέρατε στην παρέμβασή σας. Νομίζω ότι αυτή είναι μία από τις δυνατότητες και ενδεχομένω θα πρέπει να, ψάξουμε και για άλλες. Κύριε Καντέκ, είναι προφανές ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση όταν πρόκειται για την, για την ε, θεσμική αρχιτεκτονική, ε, εγώ είμαι κατά των μοντέλων. Υπάρχουν ίσως άλλες ε, δραστηριότητες όπου τα μοντέλα μπορούν να χρησιμεύσουν, αλλά όχι εδώ. Βεβαίως, το νόημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι μέσω της ποικιλία φτάνουμε στην ενότητα και η ενότητα εμπλουτίζεται από την ποικιλομορφία η βάση της συνθήκης λέει ότι η Ένωση θα πρέπει να σέβεται τον τρόπο με τον οποίο ε, γίνεται η αποκέντρωση. Είπατε ότι είναι ή η Ευρώπη των Εθνών ή η Ευρώπη των Περιφερειών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοια σαφής ε, ε, αντιπαράθεση. Εγώ είμαι υπέρ μιας εναλλακτικής Ευρώπης Τώρα δεν πρόκειται να ανοίξει μια σχετική συζήτηση εν σχέση με τον ε, φεντεραλισμό ή όχι στην Ευρώπη. Αλλά δεν μπορούμε να περιορίσουμε την ιδέα της ε, πολιτικής ένωσης που προσπαθούμε να πετύχουμε και να την ταυτίσουμε με την Ευρώπη, είτε με την Ευρώπη των εθνών, είτε με την Ευρώπη των περιφερειών. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια σωστή αναλογία εδώ. Κύριε Κόρτες Λάστρα, όσον αφορά τη στρατηγική της Λισαβόνας, η Επιτροπή μας ζήτησε να, δώσουμε, να αναφέρουμε τους δικούς μας στόχους και τις δικές μας προτάσεις και προσεγγίσεις όσον αφορά την επόμενη στρατηγική της Λισαβόνας. Θα πρέπει να πω Νομίζω στο Γκέτεμπερκ ήταν τελευταία φορά όπου συζητήσαμε το σημείο αυτό με τη Σουηδική Προεδρία και θα έχουμε τον πέμπτο εδαφικό διάλογο στην Πάλμα στις 8 Ιανουαρίου και για αυτή την ημερομηνία προετοιμάζουμε τις προτάσεις μας. Εγώ βεβαίως θα διαφυβάσω το σχετικό έγγραφο εγκαίρος, θα το γνωστοποιήσω. Πιστεύω ότι και για το μέλλον η στρατηγική της Λισαβόνας διατηρεί τη σημασία της. Ωστόσο, η κατάτμιση, ε, η τομεακή προσέγγιση, η έλλειψη συνέργειας, οι συνεργειών, νομίζω ότι είναι ορισμένες από τις αποτυχίες της, του παρελθόντος της στρατηγικής της Λισαβόνας. Για μένα είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την αποσύνδεση. Κινούμεθα από μια παραγωγική κοινωνία σε μια ε, κοινωνία πληροφοριών. Δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε το επικείμενο 8ο πρόγραμμα ανάπτυξης από την στρατηγική αυτή. Θα πρέπει να υπάρξει αυτή η διασύνδεση. Θα πρέπει να είμαστε υπέρ της δημιουργίας συνεργειών, υπέρ μιας παγκόσμιας στρατηγικής. Γιατί η μεσοπρόθεσμη έκθεση ε, το 2005 ήδη ε, απίθενε την προειδοποίηση λέγοντας ότι ποτέ δεν πρόκειται να πετύχουμε τους στόχους μας αν συνεχίσουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Θα επανέλθουμε λοιπόν με το έγγραφο, με, τις, με το κείμενο με τις προτάσεις μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας αυτό το τμήμα της συνεδρίασής μας, θα ήθελα να πω ότι είναι απολύτως σαφές ότι η Ευρώπη των πολλαπλών επιπέδων ε, ήδη υπάρχει, έχει λάβει ψάρκα. Νομίζω ότι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι η Ευρώπη είναι δυνατόν να αποκλείσει το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ε, ούτω ώστε να πετύχει του στόχου τη, νομίζω ότι θα πρέπει να δικαιολογήσουν, τα, να τεκμηριώσουν τα επιχειρήματά του. Δεν καλούμεθα εμεί να το κάνουμε. Ε, μια τέτοια Ευρώπη θα ήταν πολιτικά νόητη και ίσως και επικίνδυνη. Λοιπόν, νομίζω ότι καταλάβαμε σωστά το μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και μας μιλήσατε. Dear colleagues, we Αδελφοί, περνάμε στο 7, το οποίο δεν κάναμε χτες, για τις δημόσιες προμήθειες. Θα υπάρξει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ο κύριος Βλάσακ, ο εισηγητής, μπορείτε να ξεκινήσετε με την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μιλάμε για κάτι το καινοτόμο στην Ευρώπη. Οι εξελίξεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις δημόσιες προμήθειες έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις. Και φυσικά από πολύ παλιά όταν κάποια πόλη σαν παράδειγμα ή κάποιοι πολίτες ήθελαν να φτιάξουν κάτι, ήθελαν να χτίσουν ένα οχυρωματικό έργο ε, χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες ε, κάποιων ειδικών και γι' αυτό ακριβώς ε, έχουμε εδώ και πολύ καιρό μπροστά μας ακριβώς αυτές τις παραδόσεις θα έλεγα γύρω από τις δημόσιες συμβάσεις. Ο τομέας αυτός λοιπόν είναι ένα τομέα ο οποίο χρήζει καλύτερου ελέγχου αλλά και, και απλουστεύσεων. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τη διαφάνεια των διαδικασιών των δημοσίων προμηθειών θα πρέπει οι διαδικασίες αυτές να γίνουν απλούστερες, θα πρέπει να ελαφρύνουμε τα διοικητικά βάρη και αυτών που ζητούν τις υπηρεσίες ε, τρίτων και αυτών που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές. Τώρα, ειδικά με την χρήση των κοινοτικών χρημάτων για τέτοιου είδους δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλά διοικητικά εμπόδια. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι όταν ξεκινάει μια διαδικασία δημόσιας σύμβασης, ε, τα διάφορα στάδια παρουσιάζουν το κάθε ένα και διαφορετικούς κινδύνους. Προφανώς εδώ θα έλεγε κανείς ότι η σωστή εκπαίδευση των managers, ε, των δημοσίων υπηρεσιών ή των δήμων κτλ η ε, σωστή διαδικασία ελέγχου των, της επιμελητίας γύρω από τις συμβάσεις αυτές είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Παρ' όλα αυτά, οι κίνδυνοι παραμένουν, έχουμε να κάνουμε με τη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα και ό,τι αυτό ενέχει. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να απομακρύνουμε τα σημεία αβεβαιότητα τα οποία γεννούν αυτές οι συμβάσεις και θα πρέπει να βοηθήσουμε και τον ιδιωτικό τομέα να κατανοήσει και να κατέχει πάντα καλύτερα το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να κινηθεί. Στην Τσεχία, σαν παράδειγμα, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα σε έναν τομέα, τον τομέα της διαχείρισης ε, των λιμάτων. Και τα προβλήματα αυτά ε, συνεχίζουν να είναι πολύ σοβαρά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχουμε καταλήξει κάπου ε, σε σωστές διαδικασίες ε, προμηθειών και συμβάσεων. Υπάρχουν ε, οι υπηρεσίες κοινή ωφέλεια που εμπλέκονται, υπάρχουν οι δήμοι φυσικά που εμπλέκονται, υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες στον τομέα των μεταφορών που εμπλέκονται και υπάρχει γενικότερα μια φαιά περιοχή χωρίς ξεκάθαρες αρμοδιότητες είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε μία μορφή streamlining δηλαδή των διαδικασιών αυτών, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι δήμοι και οι κοινότητες πού και προς τα πού θα κινηθούν με ασφάλεια. Να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα, λέει η κυρία Χούμπνα, ε, είναι η πρώτη συζήτηση για από το θέμα αυτό. Δεν πρόκειται να πάρουμε καμιά απόφαση σήμερα. Η κυρία Ρούρα έχει το λόγο. Είμαι η συγγήτρια της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και γι' αυτό ήθελα να πάρω το λόγο για να διευκρινίσω ποιο είναι, τι είναι για μας σημαντικό στη δική μας Επιτροπή γιατί συντάσσουμε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας. Πρόκειται για τις δημόσιες ε, προμήθειες ως προς το εξή. Υπάρχει πλέον ε, μεγάλη, μεγάλος αριθμός διαδικασιών καταγγελιών. Ήδη από το 2007 υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Γι' αυτό έχουμε την άποψη στην Επιτροπή ότι είναι σημαντικό εδώ κάπου να καταλήξουμε και να διευκρινίσουμε ποια ακριβώς είναι η νομική βάση και ούτε ώστε να υπάρχει νομική ασφάλεια. Πρόκειται για το σύνολο της συνεργασίας μεταξύ των ε, περιφερειών. Ε, για παράδειγμα υπάρχει μια δήλωση του δικαστηρίου ότι οι επαρχίες οι περιφέρειες ε, αυτή στιγμή δεν ε, συνεργάζονται για να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες και δεν έχουν ιδιωτικά κεφάλαια να συμπεριλαμβάνουν σε αυτή τη συνεργασία, τότε μπορούν να αποφασίσουν μόνες τους ποια μορφή αποδίδουν σε, αυτή την, ε, σε αυτές τις υπηρεσίες. Ποια είναι η μορφή αυτών των υπηρεσιών. Υπάρχουν αποφάσεις για τις εταιρικές σχέσεις δημοσίου-δημοσίου και χρειάζεται προκήρυξη διαγωνισμού για να βρεθεί ο πρώτος ε, ιδιωτικός συνεργάτης, αλλά όχι ο δεύτερος. Τώρα, όσον αφορά όλα αυτά τα θέματα, είναι σημαντικό να διευκρινιστούν για να δούμε ποια είναι η νομική βάση και να υπάρξει μια επισήμανση προς την Επιτροπή, γιατί η Επιτροπή το 2010 με το Midterm Review θα ασχοληθεί με το θέμα των δημόσιων προμηθειών. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια ε, και διευκρίνηση αυτών των θεμάτων. Συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή σας και από τη δική μας πλευρά θα ήθελα να επισημανθούν οι τομείς εκείνοι οι οποίοι ε, ε, εκεί όπου έχουν συμπληρωθεί τα κενά από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και όπου υπάρχει μια ξεκάθαρη διευκρίνηση και αυτό να γίνει σαφές στις κοινότητες και τους Δήμους σε πολλούς τομείς υπάρχει το λεγόμενο soft ε, law για τα green procurements, τις πράσινες προμήθειες. Και εδώ θα πρέπει να καταλήξουμε κάπου, ώστε να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ των ε, υπηρεσιών της Επιτροπής που ασχολούνται με τις δημόσιες προμήθειες. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μία ιστοσελίδα και αυτό ισχύει και για τα κριτήρια. Υπάρχουν τα κριτήρια των οικολογικών συμβάσεων λοιπά. Εκεί θα, υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη νομική ασφάλεια. Γιατί εδώ και μήνες περιμένουμε ε, το σχετικό, τη σχετική βίβλο της Επιτροπής και αναμένουμε να εκδοθεί αυτή η βίβλος ούτως ώστε να έχουν οι Δήμοι μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά για παράδειγμα αυτές τις ε, πράσινες ε, προμήθειες. Ο Σίμων έχει το λόγο, ο Σαν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριο Ρούλε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι χρειάζεται αυτή η νομική ασφάλεια και σε, εκείνες, σε εκείνους τους τομείς που εξετάζουμε εδώ στην Επιτροπή περιφερειακή Ανάπτυξης γιατί αν δούμε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για την εκτέλεση του προπολογισμού, είναι πολύ χρήσιμο να δούμε ποια είναι τα προβλήματα για την εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων, ιδιαίτερα όσον αφορά εσφαλμένη ανάθεση έργων. Θα πρέπει να σκεφτούμε ποιε είναι οι συνέπειε στις οποίε θα πρέπει να οδηγηθούμε για να μην έχουμε ε, τέτοιου είδου ε, προβλήματα κατά την εφαρμογή όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή τα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν. Και θεωρώ, εάν δούμε τους αριθμούς, 63% ε, των ε, προγραμμάτων ε, έχουν σφάλματα, λέει έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Είναι σημαντικό λοιπόν εδώ να μην πούμε στο δημόσιο ή στους δήμους ότι έκαναν εσφαλμένα την ανάθεση αλλά πολύ συχνά, όπως υπόθηκε, ε, υπάρχει, γίνονται λάθη λόγω άγνοιας. Ε, δεν γίνονται σκεμμένα κάποια σφάλματα. Και αυτό αφορά συγκεκριμένα την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και των κονδυλίων του κοινωνικού ταμείου. Θα πρέπει να σκεφτούμε ε, ποια νομική μορφή ε, ποια, ε, τι μορφή θα πρέπει να προσλάβει η νομική ασφάλεια ούτως ώστε να μην διαπράττονται μελλοντικά αυτά τα ασφάλματα κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων του Κοινωνικού Ταμείου. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να πω κάτι σχετικά. Νομίζω ότι στο σχετικό δίκαιο υπάρχουν ε, ποικίλε διατάξεις. Και όσο και σημαντικές να είναι αυτές οι ρυθμίσεις που αφορούν τον ανταγωνισμό, την προστασία του κλίματος, την προστασία των νέων κλπ. Παρόλα αυτά, μέσω της, ε, με την πληθώρα όλων αυτών των διατάξεων του soft law κλπ, η σωστή διεκπαιρέωση των προμηθειών του δημοσίου έχει γίνει πολύ δύσκολη, ιδιαίτερα όσον αφορά του μικρούς δήμου και κοινότητε. Εκεί είναι συχνά, δεν είναι συχνά δυνατό να διεκπεραιώνει κανείς 100% σωστά αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη διαφάνεια, μια απλούστευση και μια διευκρίνηση και για τις κοινότητε και του δήμου, Έτσι λοιπόν οι εθνικές, περιφερειακές αλλά και τοπικές αρχές του δημοσίου θα έχουν ευκολότερα τη δυνατότητα να ενεργούν όσον αφορά τις ε, προμήθειες συμβατά με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και όπως είπε ο Ζήμων, ορισμένα ε, προβλήματα τα οποία προκύπτουν κατά την, ε, όσον αφορά τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου δεν είναι σφάλματα τα οποία έγιναν εσκεμμένα ή ενσυνείδητα αλλά υποκρύπτουν άγνοια όσον αφορά ε, ακριβώς αυτή την έλλειψη διαφάνειας. Γι' αυτό ο στόχος μας ε, θα πρέπει να είναι όχι να δημιουργήσουμε νέο δίκαιο, επιπλέον διατάξεις, αλλά αυτό το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή να το διαρθρώσουμε με υψηλό βαθμό διαφάνειας, ούτως να υπάρχει σωστή δυνατότητα εφαρμογής. Και μέσω αυτής της σωστής εφαρμογής και της διαφάνειας ε, να έχουμε μια πιο σωστή διάρθρωση. Αυτό δεν μπορεί να είναι ισόφελος αυτή τη επιτροπή. Ευχαριστώ. Thank you, Chair. I would like to say two... Δύο πράγματα. Σχετικά με, τα, με τις πιστώσεις. Αν δει κανείς το Περιφερειακό Ταμείο πριν από την κρίση, και τις δημοσιονομικές προοπτικές 2000-2006 διαπιστώνει ότι οι δραστηριότητες οι οποίες στρέφονται στις αστικές περιοχές για διάφορα προγράμματα έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με πολύ μικρότερα επίπεδα επάρκειας πιστώσεων από ό,τι σε άλλους τομείς. 80%, 82%, 83% και φτάνουμε στο τέλος αυτών των ε, δημοσιονομικών προοπτικών. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών όταν συζητάει τα θέματα αυτά διαπιστώνει ότι οι χώρες ζητούν χρήματα για προσπάθειες και παρεμβάσεις στο εσωτερικό των πόλεων, αλλά δεν προχωρούν στην εκτέλεση των πιστώσεων αυτών. Και δεν υπάρχει ανάλυση για το, για το γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το δεύτερο είναι κάτι το πιο συγκεκριμένο. Μιλάμε για μια ας πούμε συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οι πόλεις, οι δήμοι χρησιμοποιούν κοινοτικά χρήματα για να γίνουν πιο αποτελεσματικές ενεργειακά. Υπάρχουν πολλά προγράμματα τα οποία έχουν σαν στόχο να προσελκύσουν θα έλεγα πιστώσεις και να μονώσουν καλύτερα τις κατοικίες να ξοδεύουμε λιγότερα χρήματα από ό,τι ξοδεύουμε σήμερα για θέρμανση, σαν παράδειγμα. Τα προγράμματα αυτά δεν υπάρχουν ουσιαστικά και αυτό οφείλεται στο ότι οι μικρές κοινότητες που ελέγχουν θα έλεγα αυτές τις, ε, την κοινοτική κατοικία πρέπει να συνεισφέρουν οικονομικά. Και σήμερα οι τράπεζες δεν δίνουν ουσιαστικά δάνεια ούτε στις τοπικές αρχές και δεν παίρνουν εγγυήσει για τα δάνεια αυτά, τις κατοικίες, τις δημοτικές ή τις κοινωνικές, ανάλογα με τη χώρα. Οπότε δεν προχωρούν αυτά τα προγράμματα, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστική συγχρηματοδότηση. Οπότε οι πόλεις αναγκάζονται να κάνουν άλλα πράγματα. Να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά είτε για σχολεία, είτε για νοσοκομεία κτλ. Και ούτε και αυτό είναι εύκολο βέβαια γιατί ε, ακριβώς τα χρήματα αυτά έχουν σαν στόχο την βελτίωση της μόνωσης της ιδιωτικής κατοικίας. Πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι δηλαδή, γιατί στο τέλος δεν θα καταφέρουμε να μειώσουμε την καταναλούμενη ενέργεια. Και η κοινωνική κατοικία θα παραμείνει ενεργοβόρα. Αυτό λοιπόν το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ και δεν είναι ένα νομικό πρόβλημα, Είναι σαφές πάντως ότι τα προγράμματα αυτά τα οποία αφορούν το εσωτερικό των πόλεων, το κέντρο των πόλεων, δεν λειτουργεί σωστά και δεν υπάρχει ανάλυση για τους λόγους για τους οποίους δεν λειτουργεί σωστά. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την οικονομική κρίση. Αυτά τα ανεπαρκή αποτελέσματα τα είχαμε διαπιστώσει και πριν από την εκκίνηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οπότε διαρωτάται κανείς, θα πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια διεύθυνση την οποία ακολουθήσαμε μέχρι τώρα. Τι νόημα έχει. Υπογραμμίζω λοιπόν αυτές τις παρατηρήσεις μήπως μπορέσουμε και λύσουμε το πρόβλημα. Όλμπεχτς. Αυτό που θα πω δεν έχει και μεγάλη σχέση με τις δημόσιες προμήθειες. Πράγματι το να δώσουμε περισσότερα χρήματα στις παρεμβάσεις σε επίπεδο πόλεων ή αστικών περιοχών δεν είναι κάτι το οποίο ε, θα βοηθήσει σίγουρα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο δημοσιονομικός έλεγχος σύμφωνα με το ελεγκτικό συνέδριο καταδεικνύει ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα προκύπτουν λόγω των κρατικών προμηθειών. Μπορεί να μην σύμφωνο με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά υπάρχουν προβλήματα με τις δημόσιες προμήθειες. Και θα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η απόφαση του ΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι θέμα συμβατότητος με τη συνθήκη τα διάφορα στάδια των δημοσίων προμηθειών, η ανάθεσή τους κτλ. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο ζήτημα. Επίσης, ε, θα πρέπει να απαντήσουμε αν θα πρέπει να εναρμονίσουμε τα πάντα, όλα τα στοιχεία στα πλαίσια των δημοσίων προμηθειών μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια ή αν αντίθετα θα σταματήσουμε κάπου και θα πούμε από εδώ και πέρα, από εδώ και κάτω δηλαδή, είναι η εθνική νομοθεσία που ισχύει. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ασυμβατότητες μεταξύ της εθνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες προμήθειες και ε, της ευρωπαϊκής. Και έρχεται το ελεγκτικό συνέδριο και λέει προσοχή κύριε λάθος. Ποιος ε, ευθύνεται για το λάθος όμως. Δεν ξέρουμε. Θα ήθελα λοιπόν ο εισηγητής να εξετάσει εμβριθώς την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για να μας προτείνει τι πρέπει να αποφασίσουμε. Θα ρυθμίζουμε τα πάντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι και το σταχτοδοχείο στο γραφείο. Τέλο πάντων, σταχτοδοχείο που λέει ο λόγος ε, γιατί τώρα κάπνισμα στα γραφεία ή μήπω θα πρέπει κάποια σημεία, τα, κάποια θέματα να τα αφήσουμε στη διακριτική ευχέρεια των περιφερειών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βεσέκ ανέφερε κάποια θέματα που θα αναφέραμε όλοι. Η απλούστευση της δημοσίας προμήθειας, η αύξηση της διαφάνειας, η άρση της αβεβαιότητας και ο ανταγωνισμός. Ανέφερε ιδιαίτερα ότι οι πολλοί τοπικοί φορείς έχουν τους ε, δικούς τους ε, ε, διάβλους τροφοδοσίας, τους δικούς τους κανόνες. Εγώ πρόσφατα συνάντησα έναν συναλλασσόμενο ο οποίος υπέβαλε για να λάβει δημόσιο έργο μια πρόταση κατά 5 εκατομμύρια φτηνότερη από ανταγωνιστή του και την έχασε. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς θα πρέπει να διορθωθεί ως κατάσταση. Ο κύριος Σόμπερ Μάιρ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στην ε, προηγούμενη συζήτηση μιλήσαμε πολύ για την αποδοχή των περιφερειών αλλά και των δήμων και των κοινοτήτων. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και σχέση με αυτό που είπε ο προηγούμενος ομιλητής. Είναι σημαντικό οι κοινότητες ε, οι οποίοι εξασφαλίζουν για την ποιότητα ζωής των πολιτών ε, θα πρέπει να κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη. Και αν θέλουμε να συνεχίσουμε να μην είμαστε δημοφιλείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, αυτοί που έχουν πάρα πολλή δουλειά όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κλπ. Μιλάω για τους δήμους και τις κοινότητες, την, ε, το νερό, την ηλεκτρική ενέργεια κλπ. Όσους μεριμνούν για όλα αυτά. Αυτοί έχουν μια πολύ δύσκολη δουλειά γιατί έχουν από τη μία οικονομικά προβλήματα, από την άλλη έχουν να αντιμετωπίσουν και τι υψηλέ προσδοκίε των πολιτών. Κάτι που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο ε, το έργο τους. Γι' αυτό λοιπόν βρίσκω θετικό το να πούμε ε, να συσταθεί ένας κατάλογος ε, βασικών αρχών. Νομίζω ότι αυτό δεν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και θα ήθελα να σας πω ένα παράδειγμα. Στις κοινότητες εγώ προέρχομαι από αυτό το χώρο της κοινωτικής πολιτικής. Ε, πάντα θέλουμε να, να επιλέξουμε αυτό που κάνει την καλύτερη προσφορά. Αλλά αυτός που κάνει την καλύτερη προσφορά δεν είναι κατά ανάγκη πάντοτε και ο φτηνότερος. Ε, αυτή η σύγχυση δεν είναι πολύ λογική, αλλά γίνεται πολύ συχνά και την συναντούμε πολύ συχνά στην καθημερινή μας ζωή. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία, είναι πολύ δύσκολο να προετοιμάζεται κανείς σοβαρά για μια συνεδρίαση όταν δεν έχει στη διάθεσή του τα αντίστοιχα έγγραφα. Για παράδειγμα, χθε το μεσημέρι δεν υπήρχε κανένα έγγραφο για αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Χθε το μεσημέρι online δεν υπήρχε τίποτα. Παρακαλώ να διορθωθεί αυτό στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Δεν υπάρχουν άλλοι που θα ήθελαν το λόγο. Ένα πράγμα να πω μόνο. Έχω την αίσθηση ότι μιλάμε για μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση από πλευρά της επιτροπή μας. Και θα ήθελα όλοι οι συνάδελφοι που πήραν το λόγο και που θεωρούν ότι είναι κεφαλαιόδου σημασία στο θέμα αυτό των δημοσίων προμηθειών και ο ρόλος που έχει στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής, ο κύριος Βλάσεκ να του στείλετε, στον κύριο Βλάσεκ να του στείλετε όλα τα σχόλιά σας για να ανταλάβει υπόψη. Να υπογραμμίσω επιπλέον κάτι. Στην περίπτωση των δημοσίων προμηθειών η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής πληρώνει θα έλεγα ένα πολιτικό τίμημα άδικο. Στις περισσότερες περιπτώσεις όπου υπάρχει μια παραβίαση των νόμων για τις δημόσιες συμβάσεις Έρχονται ελεγκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ανακαλύπτουν μέσω των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής ότι η μεταφορά των ευρωπαϊκών οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις στα εθνικά συστήματα δεν γίνονται σωστά. Για πάρα πολλά χρόνια γίνεται κάτι τέτοιο. Κάποιος λοιπόν δεν κάνει σωστά τη δουλειά του για τον έλεγχο της μεταφοράς ε, των κοινοτικών ρυθμίσεων στις εθνικές ρυθμίσεις. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό έτσι, γιατί αυτό ταυτίζεται μετά με τις αδυναμίες, σαν αδυναμία μάλλον, της πολιτικής συνοχής, ενώ δεν είναι ουσιαστικά. Είναι ένα θέμα περισσότερο νομικό, ένα θέμα ρυθμιστικό, διοικητικό και επηρεάζει πολύ αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι δημόσιες συμβάσεις, ε, συνάπτονται οι δημόσιες συμβάσεις σε εθνικό επίπεδο πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η εσωτερική αγορά ελέγχεται και ελέγχει ε, τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται οι κοινοτικές ρυθμίσεις στην εθνική αρχιτεκτονική. Γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση λοιπόν θα παραμένει ανοιχτή γιατί δεν θα πρέπει να πληρώνουμε, όπως είπα, ένα ιδιαίτερα υψηλό πολιτικό τίμημα. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια λοιπόν. Θα περιμένουμε την έκθεση από πλευρά του κυρίου Βλάσεκ. Οπότε θα ήθελα... Α, θα ήθελε το λόγο ο κύριος Βλάσεκ. Ναι, θα έπρεπε να σας δώσω το λόγο. Συγγνώμη κύριε Βλάσεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι πήραν το λόγο, να πω ότι συμφωνώ με τις περισσότερες από, με όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν. Σε προσωπικό επίπεδο αυτό το οποίο ελπίζω είναι να αναλυθούν οι περισσότερες δυνατές ευθύνες σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί εκεί ε, καλούμεθα να δαπανίσουμε τις συγκεκριμένες, να εκτελέσουμε τις συγκεκριμένες πιστώσεις. Έχουμε λοιπόν συλλέξει εμπειρίες, θετικές και αρνητικές. Ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους έχουμε, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να πετύχουμε τη μείωση του διοικητικού άχθους. Περνάω στο σημείο 3. Ανακοινώσεις που αφορούν τη συνάντηση των συντονιστών χθες. Να σας ενημερώσω για τις αποφάσεις των συντονιστών λοιπόν. Πρέπει να δοθεί μια νομοθετική γνωμοδότηση για την ε, αρρωγή την προενταξιακή. Το ΕΛΚ την ανέλαβε, αναμένουμε την ανακοίνωση του ονόματος του βουλευτού. Μετά ε, για τις ακροάσεις ε, των υποψηφίων επιτρόπων. Θα θυμάστε ότι ξεκινάμε στις 11 Ιανουαρίου τη σειρά των ακροάσεων. Στα τέλη της εβδομάδας κατά πάσα πιθανότητα θα λάβει η χώρα, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Οι συντονιστές υποστήριξαν την ιδέα να υπάρξει μία ακόμα συνάντηση αυτών, των συντονιστών δηλαδή, πριν την ε, ημερομηνία της ακρόασης. Συζητήσαμε και τις μελέτες που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε την εργασία μας σε ό,τι αφορά την μελλοντική πολιτική. Συμφωνήσαμε για πέντε μελέτες, θα λάβετε τον κατάλογο. Επίσης, είπαμε, συμφωνήσαμε ότι όταν δούμε το κόστος των μελετών και το υπόλοιπο ποσό που θα έχουμε στη διάθεσή μας, θα επανέλθουμε επί της συζήτησης αυτής ε, δρυμύτερη. Επίσης, συμφωνήσαμε για τους όρους αναφοράς της Επιτροπής μας. Θα στείλω την επιστολή στον Πρόεδρο Μπουζεκ και θα σας το διαβιβάσω και σε σας μέλη της Επιτροπής αυτής, πολύ σύντομα. Επίσης, συζητήσαμε την νέα συνάντηση με τα εθνικά κοινοβούλια. Για τους νέους συναδέλφους να αναφέρω ότι η πρώτη συνάντηση ε, σε αυτά τα πλαίσια έγινε το Φεβρουάριο του 2009, φέτος δηλαδή, και συζητήσαμε το μέλλον της, της πολιτικής συνοχής. Η επόμενη έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο και θα συζητήσουμε πάλι το ίδιο θέμα, αλλά υπό το πρίσμα, εις το πλαίσιο αν θέλετε, της νέας συνθήκης. Συμφωνήσαμε επίσης να συγκαλέσουμε έκτακτη συνάντηση της Επιτροπής μας τον Οκτώβριο στα πλαίσια των ε, ε, ανοιχτών ημερών, Open Days, και ε, αυτό στις 4 Οκτωβρίου. Uh, then we also, the coordinator... Επίσης, οι συντονιστές υποστήριξαν την ιδέα να απαντήσουμε θετικά, να ανταποκριθούμε στην επιστολή Σβένσον, στην Επιτροπή μας δηλαδή να παρακαθίσει και ένα μέλος που θα επιφορτιστεί με το θέμα του gender mainstreaming. Η κυρία Σρέτερ διορίστηκε. Ισότητα των φίλων που λέγαμε παλιά, των γενών λέμε τώρα. Επίσης, ένα θέμα που είναι σημαντικό για μα, αλλά που δεν αποτελεί κομμάτι της εντολής μας είναι η ισότητα των φύλων και αποφασίσαμε ο, ο πρώτος ε, συντονιστής να διοριστεί για να παρακολουθήσει και τα θέματα που αφορούν τα προγράμματα της διασυνοριακής συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο. Ε, τώρα, κάτι άλλο, μια διάσκεψη στην οποία συμμετέσχα εγώ την περασμένη Τρίτη για να εκπροσωπήσω την Επιτροπή μας, ε, στη διάσκεψη δηλαδή της αξιολόγησης ε, της πολιτικής συνοχής. Είναι μια συνεχιζόμενη, μια τρέχουσα διαδικασία. Πριν από κάποιους μήνες ήρθε ο Επίτροπος και μας εξήγησε, μας εξέθεσε κάποια στοιχεία της αξιολόγησης αυτής. Μέχρι το 2006 όμως, ε, στη Βαρσοβία, επίσης έγινε μια διάσκεψη με 500, αυτή είναι που αναφέρω, με 500 συμμετέχοντες, έκανα και την ε, καταληκτική ομιλία στη διάσκεψη αυτή, εκπροσωπώντας ε, την Επιτροπή μας και καταδεικνύουμε ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να εμπλεκόμεθα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει όμως επίσημος τρόπος ή διάβλος αξιολόγησης ε, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτήν την ε, ευκαιρία που μας δίνεται γιατί δεν υπάρχει πολιτικό βήμα συζήτησης. Συμφωνώ λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ειδικά η Επιτροπή μας, θα, θα μπορούσε να αποτελέσει αυτό το πολιτικό βήμα συζήτησης για να συμμετάσχουμε πιο ενεργά, όχι μόνο στη συζήτηση των ε, αποτελεσμάτων, της απόδοσης της πολιτικής αυτής, αλλά και να αποτελέσουμε διάβλο επικοινωνίας, κομβικό σημείο επικοινωνίας για την αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής και βεβαίω να επηρεάσουμε και τη λήψη αποφάσεων στο μέλλον. Και ένα τελευταίο, ω αποτέλεσμα των χθεσινών συζητήσεων με τον κύριο Κλάου Κρυπ, αλλά και της σημερινής ε, παρουσίας του κυρίου Μπράντε, Πρόεδρου της Επιτροπής των Περιφερειών, θα ήθελα να σας απευθύνω μια έκκληση. Να είστε πιο ενεργοί στην Ολομέλεια μέσω της διαδικασίας ε, οφθαλμοθυρίας. Catch the eye. Ούτως ώστε να εμπλακούμε με πιο ε, ενεργό τρόπο στην ε, όλη διαδικασία για να ληφθεί υπόψη το περιφερειακό επίπεδο πιο πολύ, για να ληφθεί υπόψη η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση πιο πολύ, αλλά βεβαίως όλα αυτά δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε τώρα. Πάντως αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν θα πρέπει να εξαντλούμεθα, να αρκούμεθα αν θέλετε στην ανταλλαγή απόψεων εδώ μεταξύ μας. Όχι. Θα πρέπει να θέσουμε στο προσκήνιο τα θέματα που μας απασχολούν και στα πλαίσια των δομών και λειτουργιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή στην Ολομέλεια. Λαμπέρ. Παρακαλώ. Ναι. Μια τελευταία παρατήρηση σχετικά με την τελευταία φράση που είπατε. Αναφερθήκατε στις δραστηριότητες της Επιτροπής μας και στην παρουσία της στην Ολομέλεια. Είναι ε, σαφώς σημαντικό το θέμα της παρουσίας μας στην Ολομέλεια. Υπάρχουν όμως και οι προφορικές ερωτήσεις εδώ, μην τις ξεχνάτε, οι προφορικές ερωτήσεις ε, πολλές φορές έρχονται σε συζήτηση. Έχουμε να κάνουμε με το συγκεκριμένο θέμα μπροστά μας την πολιτική συνοχής ε, που είναι κάτι που θα μας απασχολήσει για πάρα πολύ ε, καιρό και είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία και επηρεάζει και επηρεάζεται και με πολλές άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι στην ημερήσια διάταξη πολλών ολομελιών και στον Δεκέμβριο θα υπάρξει μια συζήτηση. Έμαθα χθε, διάβασα έτσι και αλλιώς στο κείμενο του σημερινού Επιτρόπου. Υπάρχει λοιπόν και το μέσο των προφορικών ερωτήσεων. Σχετικά τώρα με τις κατευθυντήριες γραμμές, το έγγραφο για τις κατευθυντήριες γραμμές είναι μια καλή βάση για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση με την Κομισιόν. Πρέπει να είμαστε παρόντες φυσικά en mogelijkheden om plenair te doen, plenair eh, zaken te, te brengen. Overigens... Νομίζω λοιπόν ότι μια συζήτηση στην Ολομέλεια μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε και σε κάποιες άλλες βέβαια στιγμές της κοινοβουλευτική διαδικασίας να ασχοληθούμε με τις δημόσιες συμβάσεις και τις δημόσιες προμήθειες. Thank eh, Σας ευχαριστώ πολύ πάρα πολύ σύντομα για να απαντήσω σε αυτά τα οποία είπε ο Λαμπέρτ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο αρμόδιος επίτροπος έχει προετοιμάσει μια νέα διατύπωση, θα έλεγα, αυτού του προσανατολιστικού εγγράφου για την πολιτική συνοχής διευρύνοντας αυτό το οποίο είχε παρουσιάσει ήδη τον μήνα Απρίλιο. Πρόκειται όμως για ένα αναπίσημο έγγραφο, ανεπίσημο έγγραφο και όχι επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βέβαια δηλαδή, σε αυτή τη φάση μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες. Έχουμε το έγγραφο αυτό ήδη και θα το διανύμει η γραμματεία σύντομα. Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο είναι προσωπικό έγγραφο του Επιτρόπου, σαν τέτοιο χαρακτηρίζεται και δεν μπορεί να δημοσιευτεί επίσημα δημόσια. Γιατί δεν έχει εγκριθεί από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γκομάνης. Δεν ξέρω τις μελέτες συζητήσατε χθε και σε τι θέματα σταθήκατε χθε. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι γίνεται στην Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με το Ταμείο Συνοχής, τι έχει γίνει από το 2000-2006 και στη νέα περίοδο 2007-2013. Και αυτό το οποίο είναι σαφές, περιμένοντας κάποιες απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη πίεση προς τους βουλευτές να κινηθούν γρηγορότερα πιέζοντας για την για να βρεθούν περισσότερες πιστώσεις, για να προχωρήσουμε σε τομείς όπως η λεγόμενη προχρηματοδότηση, το pre-financing. Και έχουμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε χώρες γύρω από όλα αυτά. Ε, για σε τι οφείλονται όλες αυτές οι διαφορές. Είναι το πρόβλημα τα προγράμματα τα ίδια τα εθνικά. Μερικές φορές υπάρχουν ε, διαφορές πάρα πολύ σημαντικές, ένα προς τέσσερα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αποδώσουμε στην γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ε, δεν μπορεί να υπάρχουν χώρες οι οποίες να τα κάνουν πέντε φορές καλύτερα τα πράγματα από κάποιες άλλες χώρες. Εμείς πιέζουμε λοιπόν, αλλά στο τέλος δεν είμαστε σε θέση να φέρουμε εις πέρα σε αυτά για τα οποία έχουμε πιέσει. Εμείς βλέπουμε τους αριθμούς στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και αυτό είναι χρήσιμο. Αλλά το θέμα είναι να δούμε τώρα πόσο αποτελεσματικά είναι τα στοιχεία που συναποτελούν το πρόγραμμα συνοχής. Αλλά δεν διευκρινίζεται ακριβώς πού το σύστημα υποφέρει. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να μην ακολουθήσουμε μία κατεύθυνση χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει επί τόπου. Κοιτάξτε, η συζήτηση δεν θα ξεκινήσει σήμερα για μια ακόμη φορά. Αν θέλετε να έχετε μια μελέτη θα πρέπει να τη ζητάτε μέσω των συντονιστών. Για να διευκρινίσω λίγα πράγματα για τα διάφορα δεδομένα. Θα ζητήσω στο τέλος Ιανουαρίου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2008-2009 και να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει από το 2000 μέχρι το 2006, την προηγούμενη δηλαδή περίοδο. Μιλάμε, περνάμε τώρα για τις αυτόνομες ρυθμίσεις για δασμούς του κοινού δασμολογίου στην εισαγωγή βιομηχανικών προϊόντων στις περιοχές της Μαδέιρα και των Αζωρών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις μόνο για να σχολιάσω το θέμα που ανέφερε ο Πρόεδρος. Πρώτη παρατήρηση. Θα παρουσιάσω πρόταση τροπολογία σχετικά με αυτή την πρόταση πρόταση τεχνικής τροποποίησης ούτως υπήν του κειμένου που αφορά μόνο τις πρώτες ύλες, τα συστατικά και τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 2. Οι τροπολογίες αυτές ο στόχο έχουν να συμπεριληφθούν ε, σε αυτές τις ονοματολογίες κάποια προϊόντα που υπήρχαν στην παλιότερη ε, ε, πρόταση και που για ανεξήγητο λόγο εξυφανίστησαν. Δεύτερη παρατήρηση. Συζήτησα την πρόταση αυτή με τον κύριο Άλβες, τον συνάδελφο από τις Αζόρες, ο οποίος μου είπε ότι δεν έχει καμία αντίρρηση. Και τρίτο, αυτή η πρόταση τροπολογίας δεν ε, επηρεάζει καθόλου την, την απλουστευμένη διαδικασία την οποία ε, συζητούμε εφόσον το 46.2 άρθρο επιτρέπει ε, υποβολή τροπολογιών που αν εγκριθούν από τους συναδέρφους η κατάσταση, ε, η διαδικασία συνεχίζει ε, την πεπατημένη οδό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω την έγκριση της ομίγυρης για την μεταφορά μας από το 46.1 στο 46.2 άρθρο του καταστατικού. Θα στείλω τις ε, τροπολογίες σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και θα έχετε 21 μέρες για να τοποθετηθείτε. Και αν δεν τοποθετηθείτε μέχρι τότε θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Αν δεν υπάρχει άλλο σχόλιο από αυτού... Α, συγγνώμη, κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δεν είμαι αισκιώδης συζηγήτρια. Αλλά ο κύριος Άλμπερτς έπρεπε να πάει στο αεροδρόμιο και μου παρακάλεσε ε, να πω εκ μέρους του ότι συμφωνεί με τη διαδικασία αυτή. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Επίσης έχουμε την πλήρη υποστήριξη των σκιωδών. Έχουμε λοιπόν, άρα όλα είναι τέλεια. Περάμε τώρα στο σημείο 10. Ε, Η κυρία Ερμίνια Ματσόνη βρίσκεται εδώ. Ωραία. Θα σας δώσω το λόγο για να μην χάσουμε καιρό, αν θέλετε να μας κάνετε μία σύντομη εισαγωγή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω παρουσιάσει μια πρώτη πρόταση σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καταπολέμηση των απατών. Έχουμε τρία επίπεδα κριτικής εδώ και κάνουμε και κάποιες γενικές σκέψεις γύρω από το θέμα συνολικότερα. Για το 2008 λοιπόν, για το έτος 2008 φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση του επίπεδου κανονικότητας συμβατότητας. Υπάρχει επίσης και μια μείωση των δημοσιονομικών συνεπειών των παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί. Αυτό αφορά ε, τα διαφορετικά ταμεία, επαναλαμβάνω. Υπάρχει μια βελτίωση της κατάστασης, αν και έχει υπάρξει σε ονομαστικό επίπεδο αύξηση του αριθμού των παραβάσεων. Ένα δεύτερο σημείο αρνητικό αυτό είναι αυτό τα συμπεράσματα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2008 στα οποία κατέληξε το ελεγκτικό συνέδριο. 11% είναι η έλλειψη ανταπόκρισης για την πολιτική συνοχής. Υπάρχει το 18% των περιπτώσεων στις οποίες διαπιστούνται ένα σημαντικός χρόνος καθυστέρησης άνω των δύο ετών για την ανακοίνωση θα έλεγα την τελική και τα τελικά συμπεράσματα μετά από τη διαπίστωση της συγκεκριμένη παράληψης. Η αύξηση βέβαια των παραβάσεων που έχουν καταγγελθεί θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν κάτι το θετικό, γιατί αυτό δείχνει ότι οι αρχές οι οποίες ε, εμπλέκονται στον έλεγχο έχουν βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους. Από την άλλη ε, σημειώνουμε μία, ε, θα έλεγα, σοβαρή δυσλειτουργία. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να προσθέσω, μια και βρισκόμαστε στην φάση σήμερα της ε, ρύθμισης της τελικής λειτουργίας ε, για την περίοδο 2007-2013 υπάρχουν κάποια σημεία βελτίωσης και θα πρέπει η τάση αυτή η οποία πλέον έχει διαπιστωθεί να παγιωθεί και να υπάρξει συνέχιση της βελτίωσης τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα στην αιτιολογική έκθεση αν θέλετε αυτό το οποίο θα ήθελα ε, να προτείνω κυρίως προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών, είναι να προσπαθήσει να επηρεάσει ακόμα περισσότερο την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου του 2008 για τον λεγόμενο αποδεκτό ή μη κίνδυνο ή για το λεγόμενο αποδεκτό ή μη επίπεδο κινδύνου. Έχει μεγάλη σημασία στην προσπάθεια καθορισμού αυτού του ανεκτού επίπεδου θα έλεγα, να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης και στα εθνικά κράτη και σε επίπεδο κοινοτικών υπηρεσιών για να βελτιώσουν τις ελεγκτικές διαδικασίες με προοπτική την ομογενοποίηση των συστημάτων ελέγχου. Μια ομογενοποίηση που θα σμικρύνει τους χρόνους συλλογής δεδομένων, στοιχείων και τελικά τους χρόνους παρεμβάσεων στις καταγγελθήσεις παραβάσεις. Και μια τελευταία πρόταση είναι ε, της ε, περαιτέρω προσπάθειας για καλύτερο ορισμό ε, των ενιών της υποψίας για απάτη γιατί ακριβώς γύρω από τέτοιου είδους έννοιες όπως και γύρω από την έννοια του τακτισ... της κανονικής ή τακτικής ρύθμισης υπάρχουν πάρα πολλές αμφιβολίες ε, που γεννούν τελικά τις ε, διαπιστώσεις για απάτη. Σήμερα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή, θυμίζω, λέει η κυρία Χιούμπνερ. Σε μία εβδομάδα, η 10η Δεκεμβρίου, είναι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Χτες έγινε μια συζήτηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών γύρω από τη σύνδεση ανάμεσα στις απάτες, στα λάθη και στα μη τακτικά ή μη τακτά στοιχεία. Είναι σαφές ότι κάποια από τα λάθη, πολύ πιθανά, μπορεί να συνδέονται με μια προσπάθεια απάτης. Αλλά δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση. Δεν σημαίνει ότι αν έχουμε το ένα έχουμε και το άλλο. Και διευκρινίζεται στο ελεγκτικό συνέδριο ότι το 11% αφορά αποκλειστικά απάτες. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω στην εισηγήτρια πρώτον να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στις απάτες, τα μη τακτικά στοιχεία και τα λάθη. Είναι διαφορετικά πράγματα. Μπορεί και να συνδέονται, αλλά όχι ότι υποχρεωτικά συνδέονται. Μια άλλη παρατήρηση. Όταν συζητάμε για τις απάτες, και όπως είπε ένας συνάδελφος προηγουμένως, αν υπάρχει μία απάτη, πρώτον θα πρέπει να ενισχύσουμε την δυνατότητα της ΟΛΑΦ. Εμείς δεν μιλάμε για τη, στην έκθεση αυτή για την ΟΛΑΦ. Το θέμα δεν είναι το ελεγκτικό συνέδριο. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν ασχολείται με τις απάτες. Η ΟΛΑΦ ασχολείται με τις απάτες. Πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε ότι εφόσον υπάρχουν μη τακτικά στοιχεία, εφόσον υπάρχουν λάθη, είναι πολύ πιθανό, είναι μάλλον πιθανό λέει ο Όλμπριχτ, ότι δημιουργούνται οι συνθήκες που θα επιτρέψουν να υπάρξει απάτη. Αλλά εδώ πρέπει να αναφερθούμε στην ΟΛΑΦ. Κάποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να πάμε στις αστυνομικές αρχές. Όταν υπάρχει απάτη είναι ε, ε, κάτι το οποίο αφορά τις διοκτικές αρχές, αφορά την ΟΛΑΦ δεν αφορά τις υπόλοιπες διοικητικές υπηρεσίες ή το ελεγκτικό συνέδριο. Πρέπει να καταστήσουμε λοιπόν τον κανονισμό ξεκάθαρο, πρέπει οι κανόνες να γίνουν πλήρως κατανοητοί, πρέπει να υπογραμμίσουμε τα λάθη, ε, το ότι τα λάθη μάλλον και τα μη τακτικά στοιχεία μπορεί να δημιουργήσουν δυνατότητες για απάτες και αν τυχόν διαπιστώνονται κάποιες απάτες θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η ΟΛΑΦ. Όταν συζητάμε λοιπόν την προστασία των συμφερόντων των οικονομικών της κοινότητας, Πρέπει να δούμε αν αυτός ο τρόπος προστασίας είναι σωστά οργανωμένος, είναι σωστά λειτουργικός, αν η ΟΛΑΦ συμμετέχει σωστά, αν υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι επικοινωνίας με την ΟΛΑΦ. Ένα ε, τελικό σχόλιο. Για τα διαφορετικά ταμεία σε κάποιες χώρες οι διαδικασίες δεν είναι κακές, δεν υπάρχουν λάθη, δεν υπάρχει ε, πρόβλημα σοβαρό διοικητικό, υπάρχουν όμως απάτες. Όλα γίνονται καλά βέβαια. Στο τέλος όμως ε, πρέπει να παρέμβει η αστυνομία και πολλές φορές κάποιοι πηγαίνουν φυλακή. Δεν πρέπει δηλαδή τις διοικητικές αδυναμίες να τις ταυτίζουμε με τις απάτες. Πρέπει λοιπόν στην νομοδότησή μας να διευκρινίσουμε τα τρία επίπεδα λάθη, μη τακτά στοιχεία και απάτες. Τρία διαφορετικά πράγματα. Τα δύο πρώτα μπορεί να οδηγήσουν στην απάτη. Και είναι επίσης ε, ε, παρέτητο να τονίσουμε ότι θα πρέπει η ΟΛΑΦ να έχει όλες τις δυνατότητες να παρεμβαίνει το ταχύτερο δυνατόν. Γιατί αν δεν παρέμβει γρήγορα τότε δημιουργείται ένα κενό που είναι θα έλεγα πυρήνας περαιτέρω λαθών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν ε, μιλούμε για απάτη, είναι σαφές ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και αυστηροί, αλλά και δίκοι απέναντι σε όσους δουλεύουν σωστά. Όπως ε, γνωρίζετε, η ετήσια αναφορά του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών απέδειξε σχετικά με το οικονομικό έτος του 2008 στην Ολομέλεια την ε, περασμένη εβδομάδα μόλις ότι η συνοχή αποτελεί και παραμένει ο τομέας με τις πιο πολλές παρατυπίες. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης αποφαίνεται στο τρίτο σημείο ότι το υψηλό ποσοστό επιστροφής, το 11% για τα προγράμματα συνοχής, οφείλεται σε επαχθείς διοικητικές διαδικασίες. Όμως, στην ετήσια αναφορά για το 2008 το Σώμα των Ορκωτών Λογιστών μας πληροφορεί ότι ένα μεγάλο τμήμα του εκτιμόμενου ποσοστού παρατυπιών μπορεί να αποδοθεί στις ελλειπείς προϋποθέσεις και ότι οι αιτίε αυτών των παρατυπιών ήταν πρώτον προγράμματα είτε δικαιούχοι που δεν ανταποκρίνονταν στους συγκεκριμένους όρους των προδιάθεση κονδυλίων. Δεύτερον, σοβαρές παραλήψεις στο σεβασμό των κανόνων προμήθειας και τρίτον, συνυπολογισμός εξόδων τα οποία δεν καλύπτονται. Άρα μπορούμε να το δούμε και με αυτή την οπτική τα σημεία που μόλις ακούσαμε. Δεν πρέπει να θεωρηθούν, είναι σαφές αυτό, όλοι οι κανόνες ως επαχθείς. Αυτό είναι το σημείο που πρέπει να πάρουμε υπόψη μας. Για ορισμένες από αυτές τις επικίνδυνες περιοχές όπως οι παραβιάσεις των κανόνων δημόσιας προμήθειας, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να αρκείται στην ελεγκτική της δουλειά, αλλά παράλληλα να αποστείλει μια προληπτική οδηγία στα κράτη-μέλη και στις περιφερειακές διοικήσεις προφανώς για το πώς θα πρέπει να εφαρμόζονται σωστά οι σχετικοί κανόνες. Σε μια από τις απαντήσεις στις παρατηρήσεις του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών η Επιτροπή δηλώνει ότι τα περισσότερα σχέδια με υψηλό αριθμό παρατυπιών εντοπίζονται σε τρία κράτη-μέλη μόνο. Ποια είναι αυτά τα κράτη. Θα ήθελα να μάθω από την Επιτροπή ακριβώς για ποια κράτη-μέλη μιλούμε, ποιοι είναι οι λόγοι για αυτές τις ανυπάρκειες και αν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα προς αυτά τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Μια άλλη απάντηση προς, ε, από την Επιτροπή στις παρατηρήσεις του Σώματος των Αρκωτών Λογιστών μας πληροφορεί ότι οι Γενικές Διευθύνσεις για την Περιφερειακή Πολιτική και την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και τις Ίσες Ευκαιρίες έχουν δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους για την αποτελεσματική λειτουργία των διοικητικών και ελεγκτικών συστημάτων σε 545 επιχειρησιακά προγράμματα και συμπέραν ότι όπως και το 2007 έτσι και το 2008 μόνο το 31% των συστημάτων λειτουργήσε ικανοποιητικά. Υπάρχει λοιπόν, είναι σαφές αυτό, ένα σημαντικό περιθώριο για βελτιώσεις. Τέλος, ένα στοιχείο που θα έπρεπε να αναδειχθεί σε αυτή τη γνωμοδότηση που συζητάμε είναι η πρακτική βάσει της οποίας τα κράτη-μέλη αντικαθιστούσαν τις μη αποδεκτές δαπάνες που απορρίπτει η Επιτροπή με νέες δαπάνες, οι οποίες όμως ήταν επίσης μη αποδεκτές. Άρα έχουμε κάθε λόγο να προβληματιζόμαστε. Θα θέλαμε να πληροφορηθούμε από την Επιτροπή τι ποσοστό από αυτές τις μη κανονικές δαπάνες εξαιρέθηκε από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη λήξη των προγραμμάτων της περίοδου 2000-2006 αυτά και ως πληροφορίες αλλά ως και ουσιώδη στοιχεία που πρέπει να εμπλουτίσουν το συγκεκριμένο σχέδιο γνωμοδότησης που συζητούμε. Ευχαριστώ. please. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι σε σχέση με τα όσα είπε ο προηγούμενο ομιλητή, μπορούμε να τονίσουμε ότι αυτή η έκθεση πραγματικά θέτει μια σειρά ερωτημάτων και προκλήσεων για την Επιτροπή και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας πραγματικά αξιοποιούνται σωστά. Ε, και όταν λέω σωστά, ε, θα ήθελα να πω σχέση με όσο είπε και ο κύριος Όλμπριχτ. Νομίζω ότι με την ε, διατύπωση ε, των λέξεων που χρησιμοποιούμε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όχι λόγω της νομικής σημασίας των διαφόρων ενιών, αλλά λόγω των επιπτώσεων που ενδεχομένως έχουν. Η έκθεση αυτή έχει το μέλημα να εξασφαλίσει το πώς ε, εκτελούνται το, εκτελείται ο προπολογισμό και θα πρέπει να παρεμποδίσει την απάτη. Ωστόσο, διαπιστώνονται πάρα πολλέ ε, παρατυπίε. Και στην κοινή γνώμη αυτό εμφανίζεται ως εάν όλες αυτές οι παρατυπίες τελικά οφείλονται σε απάτες. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να κάνουμε αυτή την ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ των δύο ενιών. Και νομίζω ότι η συγγήτρια ε, στην προφορική της παρουσίαση δεν είπε παρκώς ότι ανησυχεί για την αύξηση των περιπτώσεων παρατυπίας. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ένδειξη ότι θα πρέπει να παρέμβουν τα λεκτικά μας συστήματα. Και θεωρώ ότι δεν είναι ρεαλιστικό να λέμε ότι πάμε προς το μηδέν όσον αφορά τη, διαπίστωση, τη δικαστική διαπίστωση παρατυπιών ή μάλλον απα, ε, απάτης. Ε, νομίζω όμως ότι η μαλλον απα απατης νομιζω αυτού του αριθμού παρατυπιών είναι σαφής ένδειξη για, την, ε, για μια παρέμβαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω παρόλα αυτά την εισηγήτρια με την οποία συμφωνώ πολύ. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να προσπαθήσει τα όσα είπαμε στη συζήτηση να τα συμπεριλάβει όσον αφορά ακριβώς αυτή την διάκριση των ενιών παρατυπίες, σφάλματα, απάτη. Γιατί αλλιώς θα μπορούσαμε να δεχθούμε στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι οι χώρες ε, μέλη ε, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Μόνο εφόσον υπάρχει αυτή η σαφήνεια μπορούν να ανταποκριθούν και να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης μεταξύ των χωρών. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Μάρκους Πίπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, μπορούμε να ορίσουμε τις έννοιες όπως θέλουμε. Αλλά η βάση την οποία μας δίνει η συγγύητα θεωρώ ότι είναι θετική καταρχήν. Και εγώ είμαι υπέρ μιας διάκρισης, αυστηρής διάκρισης, ευρωποίησης των όρων. Ωστόσο, οι παρατυπίες είναι 11% και αφορούν κυρίως τα ερευνητικά ταμεία. Αυτό είναι η αλήθεια. Και για αυτά τα 11% θα πρέπει να πούμε ότι τρεις χώρες είναι υπεύθυνε και ονομάζονται, κατονομάζονται αυτές οι τρεις χώρες. Δυστυχώς οι χώρες αυτές δεν κατονομάζονται για πρώτη φορά, αλλά έχουν, ε, έχουν κατανομαστεί κατ' επανάληψη. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα, ότι όταν τα πράγματα πηγαίνουν συστηματικά στραβά και δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε περίπλοκες κυρώσεις για τους 27, αλλά θα πρέπει να έχουμε διμερείς διαδικασία μεταξύ της Επιτροπής και των υπεύθυνων χωρών. Και θα πρέπει να έχουμε λεγκτικούς μηχανισμούς για εκείνες τις χώρες που κατ' επανάληψη διαπράττουν αυτές τις παρατυπίες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη διευθυντική πολιτική. Δηλαδή να μην τιμωρούμε όλες τις υπόλοιπες χώρες για το γεγονός ότι λίγες χώρες διαπράττουν αυτές τις παρατυπίες. Νομίζω ότι θα έπρεπε να διατυπωθεί μια, να μια πρόταση σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Όχι. Ε, επιτρέψατε μου να πάρω και εγώ το λόγο ως μέλος αυτής της Επιτροπής. Κατανοώ ότι μιλάμε για απάτη σε αυτή την έκθεση και νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι απολύτως ξεκάθαρο. Αλλά θα πρέπει επίσης να θέσουμε το ζήτημα της ποιότητας του δικαστικού συστήματος στι διάφορες χώρες. Γιατί σε ορισμένε χώρες όπου υπάρχουν απάτες, αυτό συνδέεται με τις αδυναμίες των ε, διοκτικών συστημάτων και των δικαστικών συστημάτων. Όσον αφορά την αστυνομία, νομίζω ότι θα πρέπει βεβαίως να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε διαφάνεια, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Ε, θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη διαφάνεια. Αν υπάρχει μεγάλη διαφάνεια εδώ, υπάρχουν... είναι μικρότερη πιθανότητα για απάτη. Τώρα, θα ψηφίσουμε τον Ιανουάριο την έκθεση αυτή. Αν οι συνάδελφοι θέλουν να καταθέσουν τροπολογίες, έχουν περιθώριο μία εβδομάδα μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου να το κάνουν. Θέλετε να πάρετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι από τις παρεμβάσεις που άκουσα νομίζω ότι είναι σεμβατές με την πρόταση την οποία έχω παρουσιάσει. Είναι μια πρόταση η οποία θα έλεγα έχει κάποιες, κάποιους ε, γενικούς τρόπους διατύπωσης έτσι ώστε να υποδεχθεί σωστά τα στοιχεία τα οποία θα προέλθουν από τη συζήτηση που προηγήθηκε. Δεν θα ήθελα να καθυστερήσουμε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θα επαναλάβω όμως ότι όλες οι παρεμβάσεις που έγιναν είναι συμβατές με τις δικές μου προσωπικές προθέσεις, με αυτές τις οποίες μετέφερα με γενικό κάπως τρόπο στην πρόταση που σας κάνω. Και γι' αυτό ε, θα προσπαθήσω αυτά τα ειδικά στοιχεία τα οποία εισήγαγαν οι συνάδελφοι να τα εντάξω στην πρόταση την οποία θα καταθέσω. Ευχαριστώ, θα κλείσει το θέμα. Πηγαίνουμε στο σημείο 11. Αφορώ την, αφορά συγγνώμη, την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κρέλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι υποχρεωμένη να μιλήσω για απάτες ή σφάλματα, αλλά μπορώ να μιλήσω για την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Επενδύσεων συγγνώμη ούτω ώστε να δούμε πώς ενισχύει η τράπεζα αυτή την πολιτική συνοχής. <clears throat> Με αντίστοιχες πιστώσεις. Κατ' ουσία, η μόνη αρνητική παρατήρηση που έχω στην έκθεσή μου είναι ότι η έκθεση αυτή είναι περιεκτική, αλλά δυστυχώς λέει στα πράγματα για την πολιτική συνοχής αλλά πάνω από 70% των πιστώσεων πάει στις περιοχές σύγκλησης. Και ο... οι προσπάθειες της ΕΤΕ έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια να υποστηρίξουν την πολιτική συνοχή. Και ε, ελπίζω ότι αυτό θα συνεχίσει εν ώψη της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Και η ΕΤΕ έχει απελευθερώσει περαιτέρω δισεκατομμύρια έχει θέση στη διάθεσή μας. Και θα ήθελα να πω, αυτό δεν είναι τμήμα της έκθεσης, αλλά θα ήθελα να πω ε, στην Επιτροπή, να θέσω το ερώτημα κατά πόσο δεν θα έπρεπε να προσκαλέσουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εδώ στην Επιτροπή για να μας μιλήσει πιο λεπτομεριακά και να μας ενημερώσει για την εργασία της. Στην έκθεση και πραγματικά με ενδιαφέρει το πώς λειτουργεί αυτό το Risk Sharing Financing Facility, αυτό το χρηματοδοτικό μέσο επιμερισμού των κινδύνων. Ε, ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, συμμετέχει σε αυτό, αλλά δεν έχουμε πρακτική εμπειρία. Αν είναι δυνατόν δηλαδή να προσκληθεί εδώ ένα εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να μα ενημερώσει, νομίζω ότι αυτό θα είναι ιδιαίτερο χρήσιμο. Συνολικά θεωρώ ότι οι εργασίες τους μας υποστηρίζουν σε πολλούς τομείς. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω δανείων. Εδώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ιδιαίτερος ε, ε, χρήσιμη και ωφέλιμη και θεωρώ ότι όσον αφορά ε, ε, και θεωρώ ότι αυτό αυξάνει τη δική μας πολιτική συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια σύντομη έκθεση, είναι μια για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και είναι και σύντομη, αντίστοιχα σύντομη είναι και η παρουσίασή μου. Γι' αυτό θα κλείσω εδώ. Εάν θέλουν να κάνουν κάποιες ε, προσθήκες οι συνάδελφοι, συμπληρώσεις, ε, τους παρακαλώ να το κάνουν και θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω τη δική τους εισφορά. Και σε σχέση με, τα, με όλα όσα υπόθηκαν ε, μέχρι σήμερα στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Περιμένουμε ανυπομονησία λοιπόν τα σχόλια των συναδέλφων. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ως σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚΑ, θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζω την γνωμοδότηση αυτή, νομίζω, το σχέδιο γνωμοδότηση, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ισορροπημένο κείμενο και είμαστε πολύ ευγνώμονες που η συνθήκη της ε, Λισαβόνας δίνει μεγαλύτερο εύρος στην ε, διαχείριση των ε, κινδύνων όσον αφορά τα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όλοι γνωρίζουμε ότι Υπάρχει μια μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση με εφέ ντόμινο σε όλους τους ε, τομείς. Έχουμε απόλυτες θέσεις και κλπ. Και ο λόγος είναι ότι τελμάτωσε η πραγματική οικονομία των ε, πιστώσεων. Ε, υπάρχει έλλειψη πιστώσεων, δεν μπορούν να προωθηθούν τα επιχειρηματικά προγράμματα. και υπάρχει διαφορά μεταξύ των σωστών και κακών επιχειρηματικών ε, σχεδίων. 30 δισεκατομμύρια δίνονται στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημαντικό ποσό σε περίοδους κρίσης και αυτό είναι το σημείο κλειδί. Θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να δοθούν τα κονδύλια αυτά σε τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ούτως ώστε ε, που, που, που απασχολούν, ε, που έχουν πολλές θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ανησυχώ που ορισμένε ιδιωτικέ τράπεζες χρησιμοποιούν αυτά τα κονδύλια για να φτιάξουν τα φύλλα, του συζολογισμούς τους. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε ευρεία κλίμακα. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι η εταιρική διάρθρωση της ε, τράπεζας είναι πολύ θετική γιατί δεν έχει τη δομή χορήγησης των πριμ στα στελέχη της, όπως κάνουν άλλες τράπεζες. δηλαδή εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία. 7,6 δις έχουν προβλεφθεί για τα επόμενα χρόνια, αλλά αν πράγματι θέλουμε να γίνουμε αποτελεσματικοί θα πρέπει να προβλέψουμε περισσότερα. Μέσω της καινοτομίας θα μπορέσουμε να ωφεληθούμε από αυτά τα οποία έχουμε σαν δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος να πω ότι η κυρία Κρέλ έχει σαφώς δίκιο. και τα διαφθορτικά ταμεία έχουν ήδη δημιουργήσει θα έλεγα μια εικόνα σε χώρες όπως η Πολωνία ε, αρκετά καλή. Ε, χρηματοδοτεί και διευκολύνει το τοπικό δυναμικό ιδιαίτερα σε περιοχές σχετικά απομεμακρυσμένες. Θα καταθέσω κάποιες ε, τροπολογίες μικρής εμβέλειας οι οποίες είναι συμπληρωματικές και δεν διορθώνουν ουσιαστικά τα εξαιρετικά στοιχεία που περιλαμβάνει η πρόταση ΚΡΕΛ. Να υπογραμμίσω το άρθρο 36 του κανονισμού. Υπάρχει ο κανονισμός του Συμβουλίου 1083 σχετικά με τα ταμεία, τα περιφερειακά και το Ταμείο Συνοχής. Λέγεται ότι μετά από αίτημα των κρατών μελών υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω σε σχέση με τη νομική κατά τα άλλα πρόβλεψη και βλέποντας τις δραστηριότητες ε, μέχρι τώρα των ταμείων να δούμε ε, σε ποιες περιπτώσεις ε, οι ομάδες αυτές έχουν παίξει τον ρόλο τους γιατί ξέρω ότι ορισμένες χώρες έχουν υπογράψει συμφωνίες και εννοώ το EIF, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επένδυσης, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων λειτουργεί ε, σαν σημείο προσέλκυσης ε, χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων. Εμείς λοιπόν ένα συμφέρον έχουμε. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει μια τέτοια συνεργασία, η ολοκλήρωση του προγράμματος ε, πάει καλύτερα, προχωράει καλύτερα από ότι όταν δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο και ε, σε ποιες χώρες τα πράγματα έχουν πάει καλά, σε ποιες όχι. Εν πάση περιπτώσει δώστε μας ε, περισσότερα στοιχεία ε, για να δούμε πόσο υποστηρικτικά έρχεται η τράπεζα και το ταμείο. Γιατί αν δεν τα ξέρουμε όλα αυτά, δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά, δεν μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Και είναι δύσκολο να δούμε και εμείς από δικής μας πλευράς ποιο είναι το συμφέρον μας γιατί στην περίπτωση που βλέπουμε ότι οι δυνατότητες του Ταμείου αυτού πράγματι διευκολύνουν την εκτέλεση και την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, τότε θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες αυτές περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. δεν θέλουμε να μας δείξει ακριβώς ποιοι είναι οι πελάτες της στην τράπεζα, αλλά θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες γνώσεις για την αποτελεσματικότητα της παρέμβασής τους. Ευχαριστώ κύριε Γκομάνης, δεν έχει ζητήσει άλλο το λόγο. Νομίζω ότι αυτό που είπε η Κωνσταντσα είναι πολύ σωστό. Θα πρέπει να καλέσουμε όλους τους φορείς που ασχολούνται με θέματα επενδύσεων και το EIF και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διότι τους αφορά άμεσα η πολιτική συνοχής. Όχι μόνο πίστοση που αποτελεί κονδύλιο συγχρηματοδότησης, αλλά και με τεχνική αρρωγή και υποστήριξη και με ε, παροχή τεχνικών ή οργανωτικών συμβουλών και το EPRD και, το, και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης που συμμετέχει στην πολιτική συνοχής, όλους τέλος πάντων τους φορείς. Και είναι κρίμα που λέτε ότι δεν αντανακλάτε αυτό πλήρως στην έκθεση. Μπορούμε να τους συναντήσουμε λοιπόν όλους αυτούς τους φορείς. Ευχαριστώ Κωνσταντσα. Η καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες είναι 10 Δεκεμβρίου. Θα ψηφίσουμε το θέμα αυτό στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου. Σημείο 12. Βαν Νίστελροε. Έκθεση για την εφαρμογή των συνεργειών μεταξύ έρευνας και πολιτικής ε, συνοχής και περιφερειακής πολιτικής. Λαμπέρι στο λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, είναι εν εξελίξη η εργασία αυτή. Η έκθεση είναι ένα έγγραφο εργασίας, ένα ενδιάμεσο στάδιο, το οποίο στόχο έχει να υποδείξει την κατεύθυνση, την άγουσα που θέλουμε να λάβουμε. Είναι μια εφαρμοστική έκθεση, λίγο ευρύτερη από την έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας. Μια εφαρμοστική έκθεση λοιπόν που εξετάζει πώς η φυστάμενη νομοθεσία στην Ένωση εφαρμόζεται στην πράξη. Και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να δούμε πως σχετικοί συναφείς τομείς εντάσσονται στην περιφερειακή πολιτική. Στην περίπτωση αυτή έρευνα και ανάπτυξη και κοινή αγροτική πολιτική σε σχέση με το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητος και καινοτομίας. Δεν έχουμε μπει σε λεπτομέρειες στο παρελθόν στην εξέταση αυτής της συνέργειας, αυτής της συνεργασίας. Την πρώτη φορά που παρουσιάστηκε μια τέτοια έκθεση είχε υπό το κεφάλαιο περιφέρειες της γνώσης ακροθυγός ασχοληθεί με το ζήτημα. Υπάρχει μια περιφερειακή διάσταση στα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και τώρα θα πρέπει να δούμε πώς αυτά μεταφράζονται, μεταφράστηκαν και μεταφράζονται στην πράξη και ποιες είναι οι μελλοντικές εξελίξεις. Τι με λιγενέστε με άλλα λόγια. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, οικονομία της γνώσης, ε, την ανταγωνιστικότητα κτλ. Ε, συνδέονται με αυτό το θέμα. Ευτυχώς τα πράγματα παίρνουν μια θετικότερη κατεύθυνση. Είναι πολυσχηδέστερη η σχετική πολιτική, δηλαδή περιλαμβάνει περισσότερες διαστάσεις και στοιχεία. Η συζήτηση λοιπόν που καλούμεθα να κάνουμε, η εξέταση που καλούμεθα να κάνουμε είναι πώς έχουν τα πράγματα δυνάμει του συνολικότερου πλαισίου στο οποίο κινούμεθα. Δεν θέλω να κάνω αξιολόγηση εξ αλλά στην ε, έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρονται κάποια ε, παραδείγματα, κάποιες βέλτιστες πρακτικές. Να δούμε πώς μπορούμε να διδαχθούμε από αυτά. Το θέμα είναι πώς λειτουργεί αυτή η πολιτική. Η καινοτομία αυτή αποδίδει καρπούς στην έρευνα και την ανάπτυξη στα πλαίσια των περιφερειακών πολιτικών. Η πολιτική ερεύνης, η πολιτική καινοτομίας, επαναλαμβάνω, διευκολύνει την κυκλοφορία της γνώσης. Καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς, καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Έτσι μπορούμε να αξιολογήσουμε την λεγόμενη περιφερειακή διάσταση της έρευνας και ανάπτυξης. Αυτά βεβαίως δεν προέρχονται μόνο από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και ε, το ΙΝΚΑΠ. Ε, 67% των ταπανών αφιερώνονται σε στόχους σχετικούς με τη γνώση. Προσπαθώ λοιπόν να βάλω στην εκθεσή μου στοιχεία πρακτικά. Τώρα, το πρώτο κομμάτι της έκθεσης θα είναι πιο αναλυτικό, θα εξετάζει δηλαδή το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και το επόμενο θα στρέφεται προς το μέλλον. Να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα clusters ε, που αναφύονται παντού και στο Λονδίνο και στη Γαλλία να δούμε πώς αυτό συνδέεται με τις εθνικές αρμοδιότητες, να δούμε πώς υπάρχουν άλλα κλάστερς που έχουν πιο διεθνή προσανατολισμό. Αυτά θέλω να εξετάσω στο δεύτερο κομμάτι της εκθέσεως, το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής υπό αυτό το πρίσμα για να δούμε αν έχουμε πρικοδοτήσει αυτούς με το απαραίτητο οπλοστάσιο για να δώσουμε αποτελεσματικά τη μάχη που έχουμε ως δέσμευση αναλάβει. Ατενίζουμε το μέλλον λοιπόν στο δεύτερο κομμάτι της εκθέσεως και προσπαθούμε να δούμε τα θετικά. Διαρθρωτική πολιτική, περιφερειακή πολιτική. Είναι αντικείμενα επικρίσεων πολλές φορές. Ότι δεν αποδίδουν, ότι δεν καταλήγουν στο ευκταίο αποτέλεσμα. Η πολιτική έρευνα επίσης θέλω να δώσω μια πιο πρακτική απάντηση σε αυτές τις επικρίσεις να δούμε τι γίνεται στις χώρες, στις περιφέρειες ε, με συγκεκριμένο τρόπο για να δώσουμε μια προστιθέμενη αξία, να προσδώσουμε μια προστιθέμενη αξία στις πολιτικές αυτές. Έτσι λοιπόν πάνω κάτω θα κινηθεί ο υποφαινόμενος κατά την σύνταξη της ε, εκθέσεως. Θα πρέπει να δούμε βεβαίως πώς θα συνεργαστούμε και με την Επιτροπή Ήτρε διότι είναι προφανές ότι η διαρθρωτική πολιτική, η περιφερειακή πολιτική, η έρευνα και η ανάπτυξη ε, είναι κοινή αρμοδιότητος και με την Ήτρε και ελπίζω να τα καταφέρουμε, Πρόεδρε, και με την υποστήριξή σας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι δεν θα πρέπει να συγκρίνουμε μόνο τους στόχους αλλά και τις μεθόδους. Να μου επιτρέψετε εδώ να σας θυμίσω ότι η στρατηγική της Λισαβόνας βασίστηκε στη μέθοδο της ανοιχτής συνεργασίας, δηλαδή συνδυασμός των εθνικών σενάριων η πολιτική συνοχή βασίζεται στην αναδιανεμητική μέθοδο και στον καθορισμό ποσοστώσεων που ε, ανήκουν στα κράτη-μέλη επί τη βάση του ΑΕΠ και άλλων αντίστοιχων μέσων. Η έρευνα βασίζεται στην ουσία στην ανακατανομή ακριβώς η οποία αποφασίζεται και συγκεντρώνεται στις Βρυξέλλες και με βάση επίσης και τα κριτήρια αριστείας. Οπότε οι συνέπειες σε επίπεδο εδάφους τοπικά δηλαδή ε, δεν λαμβάνονται συνήθως υπόψη. Η πολιτική συνοχής φυσικά έχει άμεση σχέση με τον τομέα της έρευνας και πολλές φορές η έρευνα έχει ε, επιπτώσεις σε επίπεδο ανάπτυξης της υπαίθρου ή και των αστικών περιοχών Συνεπώς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την ενίσχυση της έρευνας γνωρίζοντας όμως τις συνέπειες και να μην αναλύουμε μόνο την, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα, αλλά και τις μεθόδους εφαρμογής, όπως και τις επιπτώσεις που υπάρχουν. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε και να κλείσουμε εδώ τη συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Λάμπερτ για την παρουσίασή του. Ελπίζω να έχουμε στο τέλος μια καλή έκθεση. Ίσως να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον Μάρτιο, λέει ο Βανίστελ Ρόι. Καλή ιδέα. Είναι σημαντική η έκθεση πάντως αυτή και έρχεται μια στιγμή όπου όλοι έχουν στραφεί στην αναζήτηση των προτεραιοτήτων της πολιτικής συνοχής για το μέλλον. Και πρέπει να δούμε επίσης πώς συνεισφέρουμε και, στην, και στα προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επόμενο θέμα είναι τα διάφορα. Δεν ξέρω αν κάποιος θα ήθελε το λόγο, αν όχι να σας μεταφέρω μία πληροφορία. Χθε και σήμερα αναφέρθηκαν διάφοροι στο Ευρώπη 2020, το οποίο είναι διαθέσιμο πλέον στο διαδίκτυο για δημόσια διαβούλευση. Η διαβούλευση κρατάει μέχρι τις, τα μέσα Ιανουαρίου. Όσοι όμως θέλουν πράγματι να παρέμβουν και να αντιδράσουν ατομικά στην έκθεση, αν το κάνετε πριν από τα Χριστούγεννα, τότε μπορεί πράγματι να επηρεάσει το περιεχόμενο, ενώ τον Ιανουάριο ίσως να είναι λίγο αργά αλλά θα ήθελα να σας ενθαρρύνω όλους στο Europe 2020 και στην έκθεση δεν υπάρχουν ε, επίσης ε, στοιχεία για επιμέρους, ε, είναι γενικοί στόχοι τους οποίους ημεριζόμεθα και θα πρέπει να δούμε πώς η περιφερειακή πολιτική μπορεί να είναι αναπόσπαστο τμήμα των μεθόδων που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον για την επόμενη συνεδρίαση είναι η Δευτέρα και Τρίτη